Okay, Σας ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα στην ημέρησια διάταξή μας είναι η έγκριση της ημέρησιας διάταξης ως ήθιστε. Η σημερινή συνεδρία είναι υπό την αιγίδα της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την έγκριση της ημέρησιας διάταξης. Δεύτερο σημείο είναι η ανακοίνωση της Προέδρου και όπως και σε κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα επισήμως να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τους Πολωνούς βουλευτές της Επιτροπής μας και σε όλο τον πολωνικό λαό μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Σμόλενσκ το Σάββατο που όπως ξέρουμε οδήγησε στο θάνατο όχι μόνο του Προέδρου της Πολωνίας αλλά και πολλών άλλων πολιτικών, αξιωματούχων, στρατιωτικών και ηγετών της κοινωνίας. Επομένως, σε ένδειξη σεβασμού προς όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, σας ζητώ να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή. Thank you. Και τώρα προχωρούμε στο ψητό η υπήν τη σημερινη διαταξη που είναι η ακρόαση για την χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διδάγματα από την Ελλάδα, θέματα οικονομικής εποπτείας, στατιστική, πράξεις εκτός ισολογισμού και όπως ε, σας είπα είναι μια δημόσια συνεδρίαση την οποία διοργάνωσε η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά τόσο τη χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από την κατάσταση στην Ελλάδα. Η Επιτροπή μας έχει την αρμοδιότητα για τα νομισματικά και δημοσιονομικά θέματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για τις, δημοσιο... για χρηματοοικονομικές που είναι πολλές φορές το προσκήνιο της, της επικαιρότητα. Είναι χρήσιμο λοιπόν να πληροφορηθούμε για τα θέματα αυτά. Προφανώς η Επιτροπή μας έχει ένα ενισχυμένο ρόλο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε φορά που η Κομισιόν κάνει μια νομική πρόταση, νομικού χαρακτήρα πρόταση για να βελτιώσει και να εμβαθύνει την εποπτεία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμή η παρακολούθηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν υπήρξε επαρκής ικανοποιητική. Πολλά έχουν γίνει βέβαια και πολλά γίνονται και τώρα για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ενίσχυσης της παρακολούθησης του Συμφώνου Σταθερότητος θα είναι η δημόσια συζήτηση και η εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην διαβούλευση αυτή. Όπως σας είπα λοιπόν η σημερινή ακρόαση είναι τμήμα του έργου μας και περιλαμβάνει τα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να, να αντλήσουμε και το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει μια σειρά ομιλητών για το θέμα αυτό της βελτίωσης οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της αξιοπιστίας των στατιστικών και της ανθεκτικότητας των κανονισμών και των ρυθμίσεων για τις χρηματαγορές. Θα έχουμε δύο τμήματα στη σημερινή ακρόαση. Καταρχήν, στο το τρίτο τμήμα όπου περιμέναμε να είναι παρόν ο κύριος Χριστοδούλου, έχει αναβληθεί γιατί ανεκλήθη ο κύριος Χριστοδούλου για να γυρίσει στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσει επίγοντα θέματα αλλά μας τόνισε ότι είναι έτοιμο να έρθει σε μεταγενέστερη ευκαιρία ενώπιόν μας. Δεν ήταν ότι δεν ήθελε λοιπόν να παραστεί ή ότι άλλοι εκπρόσωποι δεν ήθελαν να είναι. Απλώς, όπως ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες ενέργειες οι οποίες θα γίνουν από την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίε προφανώ έχουν προτεραιότητα έναντι τη ακροασή μα. Όπω ξέρουν επίση τα τα μέλη της Επιτροπής. Είχαμε ζητήσει να έρθει ο κύριος Σαλγάδο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε σχέση με τις προτάσεις οι οποίε θα υποβληθούν προς την Ελλάδα και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια κατάλληλη ευκαιρία πριν από το καλοκαίρι για να λάβει το λόγο ενώπιόν μας. Σε επίπεδο εισαγωγής για το πρώτο τμήμα της ακρόασης μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πώς έχει τροποποιηθεί το κλίμα της οικονομικής εποπτείας και παρακολούθησης και της διακυβέρνησης και συγκεκριμένα για τις ανταλλαγές αθέτησης υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά ε, αξιόγραφα ε, από την Ελλάδα με την Goldman Sachs και επίσης οι ανταλλαγές επιτοκίων που έγιναν το 2001. Τι έχει αλλάξει έκτοτε και κατά πόσο αυτές οι ενέργειες θα το σήμερα και κατά πόσο έχουν γίνει μέτρα να αποφευχθούν τέτοιου είδου συναλλαγέ στο μέλλον. Επίση, όπω είπαμε και, όπως τονίσαμε και προ την Κομισιόν τον Ιανουάριο, φαίνεται ότι οι μηχανισμοί οι οποίοι μετατοπίζουν το χρέο εκτό ισολογισμού είναι κάτι που χρησιμοποιούνται από πολλέ χώρε. Αυτό σημαίνει ότι το χρέο βγαίνει από την εστίαση του Συμφωνίου σταθερότητα και ανάπτυξη και πρέπει να υπάρξουν τρόποι οι οποίοι θα εμποδίσουν τέτοιου είδου ρυθμίσει, οι οποίε ουσιαστικά εξαφανίζουν τμήμα του χρέους οι ομιλητές στο πρώτο τμήμα, στην πρώτη μας, ε, το πρώτο τμήμα συνεδριάσεως, ο κύριος Ρεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Βάλτε Ράντερμάχερ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της γύρω στα επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστή σε εσά. Οι ομιλητές μας θα λάβουν το λόγο για 10 λεπτά το maximum και μετά μια διαδικασία catch the eye θα υπάρξουν ερωτήματα από τα μέλη που φυσικά θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα μονάχα θέμα για να μπορέσουν να απαντήσουν με συνεκτικό και συνοπτικό τρόπο οι ομιλητές μας. Επίτροπε Ρέεν, λοιπόν, έχετε το λόγο. Let me first uh, join you, Madam President, uh, for... Καταρχήν, ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που εκφράσατε τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια σε όλα τα μέλη αυτή τη Επιτροπής, αλλά και στον λαό της Πολωνία, λόγω της φοβερή τραγωδίας που χτύπησε τη χώρα αυτή και που συγκίνησε ολόκληρη την Ευρώπη. Αισθανόμαστε τον πόνο του πολωνικού λαού. Σήμερα, σύμφωνα με τον τίτλο, θα εστιάσω την προσοχή μου στα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από την ελληνική ε, κατάσταση και τι σημαίνει αυτό για την εποπτεία. Καταρχήν, θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τις δράσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και ημερών. Καταρχήν, τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο οι συστάσει που υιοθέτησε το Συμβούλιο σε σχέση με επιπλέον μέτρα και διόρθωση του ελλείμματος της Ελλάδας ώστε να φτάσει στο στόχο του 4% μάλλον στο στόχο της μείωσης κατά 4%. Έγιναν διάφορες αποστολές εποπτείας τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό. Και εγώ ίδιος ηγήθηκα μιας αποστολής στις αρχές του Μαρτίου όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και ο, ο υποδικητής του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου. Νομίζω πως συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με την ΕΚΤ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καθώς και με την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει τώρα μπει σε πορεία ώστε να επιτύχει τον στόχο μείωσης κατά 4% φέτος, μέσα στο 2010. Αυτό είναι πολύ βασικό πριν να προχωρήσουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χώρα. Δεύτερον, γίνεται αυτή τη στιγμή η μεταρρύθμιση του ελληνικού στατιστικού συστήματος. Και επ' αυτού ο Γενικός Διευθυντής της Eurostat, κύριος Ράντερ Μάχερ, που είναι ο εμπειρογνώμονας επί των στατιστικών, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, ε, ξεκινήσαμε μια διαδικασία κατά παράβαση από πλευράς της Κομισιόν. Στη συνέχεια, ως πρώτη ενέργεια της νέας Επιτροπής ε, υιοθετήσαμε μία πρόταση που αφορά τι ελεγκτικέ αρμοδιότητες τη ε, Eurostat. Βρίσκεται τώρα υποσυζήτηση στο Συμβούλιο και βασίζομαι στην υποστήριξή σα ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νέο μέσο το οποίο χρειάζεται ε, όπως έδειξε η ελληνική υπόθεση. Και από την Κυριακή υπάρχει και ξεκάθαρη απόφαση για έναν μηχανισμό της Ευρωζώνης για συντονισμένη και υπό οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, εάν χρειαστεί, με άλλα λόγια δηλαδή, αν κινδυνέψει η οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Ποια είναι τα διδάγματα τώρα που, που θα πρέπει να αποκομίσουμε και τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Σήμερα μόλις με τους συναδέλφους στην Επιτροπή είχαμε μια πολύ καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα που είναι η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μου, οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής, έδειξαν ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και της εποπτείας των χωρών. Όπως ε, ανακοίνωσα ως υποψήφιος επίτροπος εδώ στο Κοινοβούλιο λίγο καιρό πριν, ήδη έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε, αυτό αποτελεί μια από τις βασικές μου προτεραιότητες, αν όχι την πρώτη προτεραιότητα. Είναι σαφές ότι τα πρώτα 10 χρόνια του ευρώ ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Το ευρώ έχει εξάλλου περάσει και την δοκιμασία της χειρότερης οικονομικής κρίσης ε, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, της χειρότερης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η κρίση διεύρυνε και τις γνωστές προκλήσεις για το ευρώ και τα μειονεκτήματα του ευρώ. Η μακρονομική έλλειψη ισορροπίας ε, έδειξε τα όρια της και ο αντίκτυπος είναι πολύ ε, σοβαρός. 20 χρόνια οικονομικής παγίωσης εξαλείφθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Όσο και αν αυτά υπήρξαν σημαντικά για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Διότι εν γέννη γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας για να το κάνουμε. Η ισχύουσα συνθήκη μας δίνει χώρο για να προοδεύσουμε προς την καλύτερη και χρηστότερη χρήση των οικονομικών μέσων, των και επίσης ε, μπορούμε να προβούμε σε ένα δεύτερο πακέτο αναθεωρημένης νομοθεσίας αν αυτό χρειαστεί. Και αυτό θα βασιστεί στο άρθρο 136 που προβλέπει εργαλεία και μέσα για ενισχυμένη οικονομική πολιτική εντός της Ευρωζώνης. Θα εργαστούμε επί τη βάση τριών βασικών ε, ε, τομέων, δηλαδή ο παράγοντας μεγέθυνσης, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας καθώς και η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων. Καταρχήν, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι, είναι ένα εργαλείο στεναρό, ωστόσο το πρόβλημα είναι η έλλειψη συμμόρφωσης. Για να ενισχυθεί η συμμόρφωση θα πρέπει να ενισχύσουμε το τμήμα το προληπτικό αλλά και το ανασταλτικό του συμφώνου αυτού. Διόρθωση λοιπόν έγκαιρα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει συνοχή στην Ευρωζώνη, σε όλα τα κράτη-μέλη και να είμαστε σε καλύτερη θέση ώστε να αντιμετωπίσουμε εθνικά προβλήματα. Επίσης χρειάζεται να δώσουμε νέα έμφαση στην δυναμική χρέους καθώς και τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της ε, εθνικής οικονομίας καθώς και τους εθνικούς ε, κανόνες, φορολογικούς κανόνες. Θα πρέπει να ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στις εθνικές δημοσιονομικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο λείπει για την ώρα. Θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία εποπτείας του υπερβολικού χρέους θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί και θα πρέπει να κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τους, ε, τα κράτη που επανειλημμένα ε, παραβιάζουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εφάνει σαφώ ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε και πέρα από την απλή δημοσιονομική εποπτεία. Θα πρέπει να γίνεται εποπτεία ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες καθώς και τις ανταγωνιστικές αποκλίσεις. Η μακροοικονομική ανισορροπία μπορεί να έχει πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη γενικότερα. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, Όσον αφορά έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης, ο ad hoc μηχανισμός για την οικονομική ενίσχυση, βοήθεια μάλλον προς την Ελλάδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αυτό ε, φανεί απαραίτητο. Ωστόσο, αυτό που δείχνει σαφώς η ελληνική κρίση, πως είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσης, με ισχυρά ενσωματωμένα αντικίνητρα ώστε να καθίσταται μια τέτοια κατάσταση τόσο λίγο ελκυστική, ώστε καμιά χώρα να μην θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο και αυτό το μηχανισμό. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως το τελευταίο δίχτυ ασφαλείας, το τελευταίο καταφύγιο. Αφού δηλαδή θα έχει γίνει η ενίσχυση του συμφώνου και η μακροοικονομική εποπτεία που κανονικά θα πρέπει να εμποδίζουν το να φτάσει οποιαδήποτε χώρα τόσο μακριά ώστε να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει ωστόσο να πω, όπως μάθαμε πρόσφατα, ότι ακόμα και οι χειρότερες εξελίξεις μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Τα χειρότερα σενάρια μάλλον μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικότητα και γι' αυτό καλύτερα είναι να είμαστε ασφαλείς παρά μετά να πρέπει να πληρώνουμε τα σπασμένα. Επίση, όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε ανακοίνωση τη Επιτροπή, την οποία υποβάλλουμε προ εσά και το Συμβούλιο. Και φυσικά είμαι πρόθυμο να συνεχίσουμε τη συζήτηση τόσο σήμερα όσο και σε άλλε ευκαιρίε και προσβλέπω στι δικέ σα απόψει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση της Ευρωζώνης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ράντερ Μάχερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη ανέφερε η Πρόεδρος, Είμαι ο Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο το ρόλο μου και το ρόλο της Eurostat. Η Eurostat δεν συλλέγει άμεσα και η ίδια στατιστικά δεδομένα. Η Eurostat έχει συντονιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που συναποτελείται από τη Eurostat και από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Άρα είναι συνυπεύθυνη η Eurostat με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες ε, και στα πλαίσια αυτού του συντονιστικού ρόλου εκπονεί κοινά μεθοδολογικά πρότυπα, κατοχυρώνει την ποιότητα των δεδομένων και δημοσιεύει τα ομαδοποιημένα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σχετικά με τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα το 2004 για τα δημοσιοοικονομικά, ξέρετε εξάλλου ότι είχε εκπονηθεί σχετική έκθεση τότε από την Eurostat. Ε, αυτά τα δεδομένα λοιπόν οδήγησαν σε μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος για την κατοχήρωση της ποιότητας. Έχουν ήδη εφαρμοστεί διάφορε πρωτοβουλίε όπω ο διοντολογικό κώδικα για τα στατιστικά δεδομένα, αξιολόγηση ομοτύπων των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, ε, συγκρότηση δύο συμβουλευτικών σωμάτων, ε, το Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Οικονομική Διακυβέρνηση και η αντίστοιχη Επιτροπή. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, το 2009 δημιουργήθηκε η νέα νομική βάση για πρώτη φορά για το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων. Ε, προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε αντλήσει πάρα πολλά διδάγματα από την κρίση του 2004 και 2005 και από αυτές τις συζητήσεις ε, αναβαθμίστηκε σημαντικά το σύστημα και είναι εξαιρετικά ποιοτικό το ευρωπαϊκό ε, στατιστικό σύστημα σχετικά με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα πλέον. Η Eurostat έχει διάφορα εργαλεία συγκεκριμένα για τα δεδομένα EDP και το Συμβουλευτικό Συμβούλιο έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με αυτό που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή δεν έχουμε στη διάθεσή μας ε, τόσο καλά εργαλεία όσο ε, επιθυμούσαμε. Ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε η σημασία ε, του να εκπονούνται σωστά τα επίσημα στατιστικά δεδομένα. Παρόλα αυτά υπάρχει περιορισμός δημοσιονομικών πόρων. Πέρσι με την ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση 404 σχεδιάζει ένα σύστημα ούτως ώστε να μην υπάρχει πίεση των πόρων μέσω από μια συντονισμένη και πιο παραγωγική ε, διαδικασία εκπόνησης στατιστικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Ε, θα ήθελα να στραφώ τώρα στα δεδομένα των δημοσιοοικονομικών. Στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, οι αρμοδιότητες μα ξεκίνησαν μετά τη συνθήκη του Μάστριχ που προβλέπει ότι τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα πρέπει να βασίζονται στους εθνικούς λογαριασμού και όχι στις εθνικές διαδικασίες κατάρτιση προπολογισμού. Ε, αυτό σχετίζεται με τις σχετικές αρμοδιότητες ε, ε, του ε, Συμβουλίου ε, βάσει του κανονισμού 479 που αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2005. Χρησιμοποιούμε τους εθνικούς λογαριασμούς, συγκεκριμένα τον S95 και τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Τονίζω ότι η Eurostat ασχολείται μόνο με τα γεγονότα, τα δεδομένα που ανήκουν στο παρελθόν, αυτά που έχουν ήδη συμβεί. Ε, δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο ως προς τις δημοσιοοικονομικές προβλέψεις. Ε, ε, ο ΕΣΑ 95 προβλέπει λοιπόν ε, ειδικού κανόνες και μπορεί να προκύψουν άλλες εξελίξεις. Παραδείγματο χάρη, οι κυβερνήσεις να κάνουν άλλου είδους ε, εμπορικές συναλλαγέ. Ε, εμείς είμαστε αρμόδιοι για μια προϊούσα διαδικασία λήψη αποφάσεων και εκπόνησης μεθοδολογικών εργαλείων, ούτω ώστε να αναβαθμίσουμε την εναρμόνιση των εθνικών στατιστικών δομένων για του εθνικού λογαριασμού. Την τελευταία δέκα ετία τα, οι κυβερνήσει χρησιμοποιούν όλο ένα και πιο περίπλοκα εργαλεία λογιστική καταγραφή, οπότε από τεχνική και τεχνολογική άποψη ε, αντιμετωπίζουμε όλο ένα και μεγαλύτερε προκλήσει. Αυτά τα εργαλεία τα αντιγράφει μία χώρα από την άλλη και άρα ε, δεν πρόκειται μόνο για στατιστικολόγους που ασχολούνται μόνο με ε, καθοδηγητικές γραμμές για την εξέταση στατιστικών δεδομένων. Η Eurostat έχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Να σας δώσω ε, ένα παράδειγμα ε, μόνο δηλαδή ότι χρειαζόμαστε νέα εργαλεία ώστε οι στατιστικολόγοι να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Το 2005 για τα δεδομένα EDP ε, οδήγησε σε επίσπευση του έργου μας. Τώρα τακτικά επισκεπτόμαστε όλες τις χώρες ε, και ε, ήδη έχουμε βρεθεί στην Ελλάδα για αυτές τις μεθοδολογικές επισκέψεις και τονίζω ότι τέτοιες επισκέψεις έγιναν μόνο στην Ελλάδα για να ε, αυξήσουμε τη διαφάνεια των εργασιών μας και αυτό καταδεικνύεται από τα δημοσιοποιημένα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Αυτά για το ιστορικό υπόβαθρο και τώρα θα περάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα που μας απασχολεί. Στις 8 Ιανουαρίου του 2010 εκδώσαμε μία έκθεση για τα στατιστικά δεδομένα για το υπερβολικό έλλειμμα όπου τονίσαμε ε, τα προβλήματα που υπήρχαν σε σχέση με τα δεδομένα EDP για το 2009 ε, έγιναν σημαντικές αναθεωρήσεις ε, για τα δεδομένα ελλείμματος του 2008 από την ελληνική κυβέρνηση και το χρέος πέρασε στο 7,5% εντοπίσαμε σοβαρές ε, παρατυπίες ε, στην ε, κοινοποίηση του Απριλίου και του Οκτωβρίου του 2009 για τα δεδομένα EDP και οι αναθεωρήσεις οφείλονταν σε θεσμικές ελλείψεις στην Ελλάδα ούτως ώστε να εκπονηθούν σωστά τα δεδομένα σχετικά με το έλλειμμα. Δεν υπήρχε επαρκής διακυβέρνηση, ανεπαρκής επιμερισμός των ευθυνών ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία δεν ήταν γνωστό ποιος ακριβώς ήταν υπόλογος ε, και γενικότερα υπήρχε σοβαρή έλλειψη γραπτών εντολών από πλευράς της ε, κυβέρνησης. Επίσης, ε, ανακαλύψαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διάφορα παράγωγα για να κρύψει την αύξηση ε, του δημοσίου χρέους της ε, και μετά την έκθεση της Eurostat και την έκθεση των εξαρτήνων εμπειρογνωμόνων για την Ελλάδα προέκυψαν διάφορες συστάσεις και δράσεις παρακολούθησης και ζητήσαμε πάρα πολλές πληροφορίες από την Ελλάδα και κάναμε διάφορες επισκέψεις τον Μάρτιο του 2010. Ε, σχετικά τώρα με τη διαδικασία κοινοποίηση των δεδομένων EDP συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ούτως ώστε στο μέλλον να συγκροτηθεί ένα ε, κρατεό ε, στατιστικό σύστημα. Όπως είπε ο κύριος Όλη Ρένε, έχει κινηθεί διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή έχει εκδώσει η αναθέωση του κανονισμού 479 ε, ούτως ώστε να αναλάβει ελεγκτικές ε, αρμοδιότητες η Eurostat. Αυτή η πρόταση ε, ανοίγει νέα δυνατότητα για τη Eurostat. Δηλαδή θα έχει πρόσβαση σε σημαντικές πηγές πληροφοριών. Όπως παραδείγμα χάρη θα έχει πρόσβαση στους εθνικούς λογαριασμούς. Ε, είναι μια μινιμαλιστική προσέγγιση αυτή η πρόταση. Δεν τροποποιεί άρδιν το κανονισμό 479. Πλην όμως σε έκτακτες και σαφώς προσδιορισμένες περιστάσεις αποδίδει ελεγκτικές αρμοδιότητες για τους εθνικούς λογαριασμούς και ελέγχου των δεδομένων βάση ε, των ε, υφισταμένων μεθοδολογικών εργαλείων και ε, αυτά τα λέω για να σα περιγράψω τι είδου ελεγκτικέ αρμοδιότητε θα έχει η Eurostat. Αν εγκριθεί αυτή η πρόταση αναθεώρηση, ε, θα ενισχυθεί ε, σημαντικά η εργασία τη Eurostat ω προ τα δεδομένα EDP με εσωτερική αναδίπλωση. Και έτσι τακτικά θα μπορούν να γίνονται επισκέψει για τα δεδομένα EDP σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι ενισχυμένε αρμοδιότητε βέβαια που ζητούνται δεν ε, απαλήφουν τον κίνδυνο η θελημένης ε, ε, πλημελούς καταγραφής των δεδομένων. Μειώνουν απλώς τον κίνδυνο και όλα εξαρτώνται από το προσωπικό, από τις αρμοδιότητες και από τους πόρους που έχουν και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες φυσικά για να έχουμε σωστή λογιστική καταγραφή. Και ξανατονίζω το θέμα των πόρων. Ε, το όραμα για την Ευρωπαϊκή ε, Συλλογή Στατιστικών Δεδομένων εστιασμένο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ε, αποσκοπεί στην αύξηση των πόρων για να καλυφθούν οι τομείς προτεραιότητες. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνοδεύει τη αύξηση των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αύξηση πόρων σε εθνικό επίπεδο. Ε, ποια είναι η γενική εικόνα. Η ε, εθνική στατιστικολόγοι ε, αποσκοπούν επίσης ε, στην ε, πιθανή χρήση διαφανούς συστήματος λογιστικής καταγραφής ούτως ώστε να είναι ακέραιες οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Επίσης αναθεωρούμε τώρα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, το ΟΕΣΑ 95 θα μετονομαστεί ΕΣΑ 2010 και πολύ συγκεκριμένα για τα κυβερνητικά δεδομένα και θα γίνει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφέτος για νέο κανονισμό για να ακολουθηθεί νέα προσέγγιση για τα δεδομένα μέχρι το 2014. Ε, προπαρασκευαστικά λαμβάνουμε υπόψη όλη την εμπειρία που αντλήσαμε από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. μπορώ να πω στα μέλη ότι και τους ε, ομιλητές μας ότι θα έχουμε καταρχήν και τα γραπτά αντίγραφα των ομιλιών τους. Είναι λοιπόν καλύτερα να πούνε ποιοι δεν θέλουν να λάβουν το λόγο γιατί φαίνεται ότι όλοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβω ομαδών τις ερωτήσεις σας γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τελειώσουμε. Καταρχήν, δίνω το λόγο στην κυρία Κράτσα. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό και μόνο ένα ερώτημα. Σας παρακαλώ μόνο για ένα θέμα, ένα ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ο, κύριος Ράντερ Μάγερ μόλις μας είπε ότι η Eurostat με τις δύο εκθέσεις της το 2004 και το 2010 τον Ιανουάριο ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα που κανείς δεν αμφισβητεί της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην συλλογή δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων ωστόσο η ευρωπαϊκή επιτροπή έκλεισε το 2007 τη διαδικασία επίπαραβάση που είχε ξεκινήσει το 2004 κατόπιν των βελτιώσεων που ε, είχαν καταγραφεί από την ε, διακυβέρνηση του 2004 2005 Σε τι συμπεράσματα κατέληξε η Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των swaps από την ελληνική κυβέρνηση το 2001 αλλά και την αλλαγή του έτους καταγραφής των νοσοκομιακών δαπανών και προμηθειών στον προϋπολογισμό που είναι δομικό στοιχείο για την καταγραφή του ελλείμματος, τα οποία συνέβαλαν και σημαντικά στην αναθεώρηση προς τα πάνω των ελλημάτων. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα που ήδη μας ανακοινώσατε και αναθεώρησης είναι αρκετά για να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η αξιοπιστία των δεδομένων τα οποία θα συλλέγεται και για να μπει σε μια τάξη και η καταγραφή ε, σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ η Σόφη Ιντφέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο και τον κύριο Ράτερ Μάχερ. Το πρώτο μου ερώτημα Θέλω να πω ότι χαιρετίζω τις καλές προθέσεις και τη Κομισιόν και τη Eurostat να γίνουν πιο σφιχτοί και αυστηροί κανόνες. Μήπως όμως το πρόβλημα είναι ότι τελικά δεν θα έχουμε τα εργαλεία εφαρμογής και αστυνόμευση. Έχουμε σαφεί κανόνε στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί είναι ουσιαστικά μια συμφωνία κυρίων που επιτάσσει ότι δεν μπορεί να παρέμβει ένα κράτο μέλο σε ένα άλλο. Δηλαδή, λέει ο καθένα, εάν δεν παρέμβετε στο δικό μου χώρο, δεν θα παρέμβω στο δικό σα. Μήπω θα πρέπει όλα αυτά να είναι νομικά δεσμευτικά σε επίπεδο συμφώνη σταθερότητα. Δεύτερον, όλοι θέλουμε να δακτυλοδεικτούμε την Ελλάδα. Και ελπίζουμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμω δεν είναι μονάχα η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα σύμπτωμα μια ασθένεια γενικότερη, ενό αδύναμου συστήματο. Και θα έπρεπε να υπάρχει μια έρευνα για το κατά πόσο ήξερε η Eurostat και η Κομισιόν τι ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα και τι κάνανε και ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος των κρατών μέλων γιατί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ήταν διστακτικά να επιτρέψουν να γίνουν λογιστική έλεγχοι στους εθνικούς λογαριασμούς. Και θα ήθελα να προτείνω εδώ να γίνει μια έρευνα, ακόμα και μια εξεταστική επιτροπή για το σύστημα αυτό και το τελευταίο μου ερώτημα προς την Κομισιόν αν δω πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς που εξαπατούν στις επιχειρήσεις, όπως παραγωγικά στην περίπτωση της ΕΡΟΝ, πηγαίνουν φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως υπήρξαν και εγκληματικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περίπτωση, άτομα τα οποία επίτηδες υπενόμευσαν τη σταθερότητα του ευρώ. Ωραία λέει η πρόεδρος. Σόφι, ναι, αλλά έδωσε ένα κακό παράδειγμα, έκανε δύο ερωτήματα. Ίσως πρέπει να σου ε, επιβάλλουν ένα πρόστιμο αργότερα. Ο κύριος Έπινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η περίπτωση της Ελλάδος καταδεικνύει σαφώς ότι όταν ξεφύγει από τον έλεγχο ένας δημόσιος τομέας είναι πολύ δύσκολο να τον χαλιναγωγήσει κανείς και πάλι. Γιατί η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά εκτός των κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το μεγαλύτερο χρόνο που συμμετείχε στη ζώνη του ευρώ. Το ερώτημά μου είναι πότε θα Πότε ήξερε η Κομισιόν για το σοβαρό αυτό πρόβλημα και πότε σταμάτησε να γνωρίζει τι γινόταν. Υπήρξε πολλή χρόνος μέχρι να υπάρξει αντίθεση. Και τώρα, για τα θέματα συμμόρφωση, η κυρία Μέρκελ είπε ότι αν μια χώρα κατά συρροή παραβιάζει τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, τότε πρέπει να αποσυρθεί από τη χώρα από το χώρο του ευρώ. Υπάρχει λοιπόν στρατηγική εξόδου. Θα είναι αυτό μια πραγματική επιλογή. Μήπω θα είναι αυτό το καλύτερο αντικίνητο για μια χώρα που θέλει να κάνει τέτοιου είδους ενέργειες. Κάποιες ερωτήσει τώρα σε αυτά τα τρία ερωτήματα. Κύριε Πίτροπε, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να ξεκινήσω εγώ και μετά ο Βάλτερ Ράντεμάχερ μπορεί να συμπληρώσει αυτά τα οποία λέω σε σχέση με το ρόλο της Eurostat. Ξεκινώ με το ερώτημα της κυρίας Κράτσα σε σχέση με, τα, με τις ανταλλαγές και το ρόλο που έπαιξαν σε αυτή τη διαδικασία. Τα swaps δηλαδή. Εγώ όταν αναδύθη αυτό το θέμα ζήτησα από τις υπηρεσίες μου και την Γενική Διεύθυνση για τα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά Θέματα, την ΕΚΦΗΝ και τη Γεροστάτ να ερευνήσουν ενδελεχώς αυτή την κατάσταση. Είναι σαφές ότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κυβερνήσεις έχουν διορθώσει τα στοιχεία τους βάσει των κανόνων οι οποίοι ενεκρίθησαν το 2008 Υπήρξε λοιπόν αυτή η αναθεώρηση των κανόνων μας το 2008 και χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πολωνία διόρθωσαν τα στοιχεία τους του 2001 και άλλων ετών αναδρομικά. Η Ελλάδα όμως είναι η μόνη χώρα η οποία ακόμα δεν έχει διορθώσει τα στοιχεία ελλείμματός της, αντιστοίχως με τους κανόνες αυτούς. Αλλά επειδή ανησυχώ ιδιαίτερα από την ε, ενδεχόμενη χρήση χρηματοοικονομικών παραγόγων και ανταλλαγών αθέτησης ε, υποχρεώσεων swaps δηλαδή, για να τροποποιηθούν τα κρατικά στοιχεία και οι εθνικοί λογαριασμοί σε σχέση με το έλλειμμα και το χρέος, ζήτησα από την Eurostat να προχωρήσει σε μια σε βάθος έρευνα σε σχέση με τη χρήση εργαλείων εκτός αγοράς από την ε, από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό συζητήθηκε και από τον κύριο Ράντε Μάχερ, ίσως να πει κάτι για το θέμα αυτό. Για μένα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί το ταχύτερο δυνατό και αυτό φυσικά θα απαιτήσει την πλήρη συνεργασία των ελληνικών αρχών. Για τα ερωτήματα τώρα της κυρίας Ιντφελτ σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς εφαρμογής του Συμφωνίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια. Υπάρχουν προφανείς αδυναμίες στο σύστημα εφαρμογής και επιβολής του Συμφώνου αυτού Σταθερότητας και από πολλές απόψεις συμφωνώ ότι η πίεση των ομοτήμων απουσίαζε στην περίπτωση αυτή. Αυτά που είναι το 2003, 2004, 2005 είναι ότι κάποια κράτη-μέλη ουσιαστικά κάνανε μια συμφωνία μεταξύ τους η οποία παρέκαμψε την, τον έλεγχο της Κομισιόν και με τον τρόπο αυτό υπήρξε μια αποδυνάμωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Τώρα χρειάζεται, όχι, αν όχι να αναθεωρήσουμε, τουλάχιστον να ενισχύσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Όπως εξήγησα, έχουμε κάποια εργαλεία, Παραδείγματο χάρη βάσει του άρθρου 136 λαμβάνονται οι αποφάσει στην Ευρωομάδα από του Υπουργού Οικονομικών με παρουσία τη Κομισιόν και τη Κεντρική Τράπεζα. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται από τους υπουργού της ζώνης του ευρώ με ειδική πλειοψηφία και η χώρα η οποία εξετάζεται δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Αυτό είναι ένα καινοτόμο στοιχείο και αυτό νομίζω θα μπορέσει να εξασφαλίσει καλύτερη πειθαρχία σε ό,τι αφορά την επιβολή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, πέραν των στοιχείων τα οποία προανέφερα. Συμφωνώ τώρα ότι θα πρέπει να ρωτήσετε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη γιατί δεν υποστήριξαν τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Εγώ έχω μία απάντηση τώρα από την αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου και τώρα φαίνεται αυτό ότι είναι ελπιδοφόρο γιατί κάποια μεγάλα κρατημέλη έχουν τροποποιήσει τη θέση τους και εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα αυτό παροχής λογιστικών στοιχείων για να υπάρξουν και ισχυρότερες <clears throat> αρμοδιότητες ελέγχου στα κρατημέλη. Ο κύριος Έπινγκ αναφέρθηκε στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Εγώ είμαι στο αξίωμα αυτό από τις 9 Φεβρουαρίου του 2010. Έκτοτε έχω χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου να αντιμετωπίζω την περίπτωση της Ελλάδος και έχω λειτουργήσει φυσικά επί τη βάση των πληροφοριών που λάβαμε αμέσως και νομίζω ότι τώρα μπορώ να θεωρήσω ότι έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο, έχουμε την κατάλληλη εργαλειοθήκη μέτρων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και εξάλλου ξέρουμε ότι και η Ελλάδα έχει αναλάβει δράση για να μπορέσει να υπάρξει η μείωση του ελλείμματος στο δημοσιο τομέα. Δίνω το λόγο τώρα στον Βάλτερ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω με το θέμα αυτό της, όπως είπε ο κύριος Ρεν, του της νομικής εργαλειοθήκης η οποία πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα αυτό. Ξεκινάμε το ερώτημα της κυρίας Κράτσα. Γιατί σταματήσαμε τη διαδικασία επί παραβάση την τελευταία φορά. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πού θα υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Την τελευταία φορά η διαδικασία επί παραβάση συνεδέωτο με τις δυνατότητε ελέγχου της Eurostat, οι οποίες ήταν περιορισμένες στον λεγόμενο στατιστικό τομέα. Δεν είχαμε το 2005 λοιπόν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε πρώτερο επίπεδο και να ελέγξουμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον δημόσιο τομέα εν γέννη προς την Eurostat. Η πρώτη λοιπόν διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδος περιοριζόταν σαφώς σε δράσεις οι οποίες έπρεπε να λάβουν χώρα στην Ελλάδα σε σχέση με τον πυρήνα των υπολογισμών μηχανογράφηση στοιχείων. Έπρεπε λοιπόν να σταματήσουμε τη διαδικασία επί παραβάση όταν διαπιστώσαμε ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος έχει εφαρμόσει το σύστημα αυτό μηχανογράφησης το οποίο του ζητήσαμε να εφαρμόσουν. Αυτό το οποίο είναι διαφορετικό όμως σήμερα είναι ότι από νομική έποψη έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία επί παραβάση η οποία δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο θέμα της εφαρμογής μεθοδολογικών κανόνων στον τομέα των στατιστικών. Έχουμε ξεκινήσει όμως μια διαδικασία η οποία αφορά και την χρήση στατιστικών αρχών που είναι η αξιοπιστία των δεδομένων, η ανεξαρτησία της υπηρεσίας αυτής. Υπάρχουν λοιπόν θεσμικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόσφατη προσφυγή επί παραβάση. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί αυτές οι αρχές εδράζονται στο νέο κανονισμό για τη στατιστική 223 του 2009. Μια δεύτερη αλλαγή θα προκύψει εφόσον και όταν αναλάβει η Eurostat εξουσίες λογιστικού ελέγχου, τότε έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πριν από τα στατιστικά στοιχεία και ουσιαστικά να ανοίξουμε τα ντουλάπια και τους φοριαμούς σε διάφορες υπηρεσίες του εθνικού, ελληνικού κράτους, όπως παραδείγματος αυτό που αναφέρατε για τα νοσοκομεία. Έχουμε λάβει πολλά στοιχεία από την έρευνά μας στην Ελλάδα που δείχνουν ότι πραγματικά υπάρχει μια αλλαγή στο κλίμα, μια αλλαγή νοοτροπίας η οποία οφείλεται και στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Για τις ενδεχόμενες εγκληματικές ενέργειες πρέπει να τονίσω ότι στην πρότασή μας για τροποποίηση του κανονισμού 479 έχουμε συμπεριλάβει και μία πρόταση η οποία ζητά από τα κράτη-μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αξιωματούχοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παράδοση των σχετικών στοιχείων στην Κομισιόν κτλ. κτλ ότι θα είναι υπόλογοι και ότι θα δρουν βάσει των αρχών οι οι οποίες αρχές θεσπίζονται από τον κανονισμό αυτό, τον αναθεωρημένο 479. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικού χαρακτήρα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανακοινώσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2011 τα μέτρα αυτά στην Κομισιόν κτλ. Ο στόχος λοιπόν αυτής της αναθεώρησης είναι όχι μόνο να γίνουν πιο ανεξάρτητα και εύρωστα τα στατιστικά συστήματα, αλλά να γίνουν και υπόλογοι και να λογοδοτούν οι αξιωματούχοι από τις στατιστικές υπηρεσίες και να υπάρχει απαραίτητη ακεραιότητα και να εξασφαλίσουν τα κράτη-μέλη και να μας δίδουν σχετική έκθεση για το πώς βελτιώνουν τα συστήματα αυτά σχετικά. Επομένως, αυτό περιλαμβάνεται μέσα στην πρότασή μας για τον αναθεωρημένο κανονισμό. Τελευταίο και όχι ίστατο θέλω να αναφέρω ότι ό,τι και να κάνουμε μέσα στη νομική εργαλειοθήκη για τη βελτίωση αυτής της εργαλειοθήκης δεν θα ευδοκιμήσει η προσπάθειά μας όσο είναι αδύναμες οι στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι εύρωστες σε ό,τι αφορά τους πόρους και ανεξάρτητες. Και θέλω και πάλι να υπενθυμίσω ότι η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος η συνεργασία μας λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα μπορεί να μας επιτρέψει να έχουμε ανακατονομή των πόρων. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν πρόσθετοι πόροι, απλώς χρειάζεται περισσότερη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα τόσους πολλούς που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις που θα ακούσουμε πέντε στον επόμενο γύρο. Ούντο Μπούλμαν η Άννη Ποδηματά, ο κ. Ε, Χωζέ Καρσία Μαρκάλιο. Και θα ακούσουμε πρώτα τον Ούντο Μπούλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Ράντε Μάχα. Στην ανάλυση που παρουσιάσατε για αυτά τα οποία έγιναν, θα ήθελα να σταθώ εκεί και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Ρεν για το τι θα γίνει στο μέλλον όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Κύριε Ράντεμαχερ, ένα ερώτημα μετά από την δήλωση που κάνετε τώρα για την ε, αλλαγή της νομικής κατάστασης, την αλλαγή της νομικής βάσης επί της οποίας μπορείτε να λειτουργήσετε. Τι ίσχυε όταν ξεκίνησαν οι πράξεις με, με τα χρηματοοικονομικά παράγοντα. Παράγωγα. Υπήρχε η υποχρέωση Δήλωση από, την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε, είχατε γνώση για το θέμα αυτό ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία με την Goldman Sachs και δεχομένως και με άλλους χρηματοοικονομικούς ήχου σε σχέση με συναλλαγέ για παράγωγα. Γνωρίζατε ότι ίσως άλλα κράτη-μέλη κάνανε χρήση τέτοιων εργαλείων ή χρησιμοποιούν ακόμα. Αυτό θα μας ενδιέφερε. Προφανώ υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να συζητήσει κανεί για το ελληνικό παράδειγμα και τώρα στρέφομαι στον κύριο Ρέν για το επόμενο ερώτημα. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό στην περίπτωση της Ελλάδος είναι ότι υπάρχει κερδοσκοπία κατά κρατών μελών και κερδοσκοπία κατά του ίδιου αυτού του ευρώ. Η δική μου άποψη και η άποψη της ομάδας μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να αναχαιτήσουν την κερδοσκοπία κατά του ευρώ και να εξασφαλίσουμε στο μέλλον μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούνται σε λογικές συνθήκες οι οποίες δεν υπόκεινται στη δράση των κερδοσκόπων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά που έγινε το Σαββατοκύριακο είναι πραγματικά ένα βήμα προς τα εμπρός. Μια ακόμα πιο ευρωπαϊκή λύση θα ήταν ακόμα καλύτερα. Μια λύση όπως αυτή που χρησιμοποίησαμε στην περίπτωση χωρών ε, που δεν ήταν μέλη της Ευρωζώνης βάσει του άρθρου 153. Θεωρείτε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας τέτοια διαδικασίας η οποία θα μπορέσει να δώσει ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό για να αντιμετωπίζει τέτοιες κρίσεις στο μέλλον ή όχι. Η Ανυποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πολύ σύντομα κύριε Ράγκεντερ Μάρκετ. Νομίζω ότι πρόκειται περί λάθος της διερμηνίας αλλά θα ήθελα να μα διευκρινίσετε, επειδή εμφανιστήκατε να λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί στον Ενεστώτα παράγωγα ε, για να κρύψει το χρέο τη, ότι προφανώ αυτό είναι λάθο και ότι αναφέρεστε στο παρελθόν. Ε, κύριε Επίτροπε, σε ό,τι αφορά τον ε, μηχανισμό στήριξη οικονομιών με μεγάλε με μεγάλες δυσκολίε όπω η Ελλάδα στην προκείμενη περίπτωση, συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για μια καθοριστική σημασία απόφαση και για την ελλάδα και για την ευρώπη. θέλουμε να πιστεύουμε ότι δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας και για το ευρώ και για την ελληνική οικονομία όμως ε, βλέπουμε ότι ακόμα και μετά από την σημαντική απόφαση του eurogroup της κυριακής που αποσαφηνίστηκε σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του μηχανισμού και υπήρξε ένας πρώτος θετικός αντίκτυπος στις αγορές την επόμενη μέρα βλέπουμε σήμερα από σήμερα μάλλον να επιστρέφει σιγά σιγά στο προσκήνιο μια κακοφωνία αντικρουόμενες δηλώσεις σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης και εφαρμογής αυτού του μηχανισμού και επειδή αυτές οι αντικρουόμενες δηλώσεις και η κακοφωνία ήταν εξ αρχής το μεγάλο μας πρόβλημα και υπονομεύουν και τη σταθερότητα του ευρώ και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον ελληνικό λαό κυρίως για να εξηγιανθεί η ελληνική οικονομία και για να περισταλεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω, εξακολουθούν να υπάρχουν ασάφειες γύρω από τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού και αν ναι, μέχρι πότε θα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ασάφειες. Μένουν ακόμα ζητήματα προς διευθέτηση. Εάν δεν υπάρχουν ακόμα ασάφειες, κύριε Επίτροπε, με ποιο τρόπο θα σταματήσει, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτού του είδους τις δηλώσεις κακοφωνίας που υπονομεύουν στην πραγματικότητα απριόρι την αποτελεσματικότητα αυτού καθεαυτού του μηχανισμού στήριξης που αποφασίσαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, λέγεται ότι οι οικονομολόγοι είναι οι καλύτεροι προφήτες, αλλά για το παρελθόν μονάχα. Εγώ νομίζω ότι για μια φορά πρέπει να μιλήσουμε καλύτερα για το μέλλον. Θα ήθελα να μου πείτε κύριε Επίτροπε και ο, αρμόδιος για τη Eurostat, ο διοικητής διευθυντής Ευρωστάτ, αν έχουμε ξεκινήσει να παίρνουμε μέτρα για να ποσοτικοποιήσουμε τις υποχρεώσεις εκτός προϋπολογισμού που προφανώς βαρύνουν τα κράτη-μέλη και τα υποχρεώνουν να εξηγιάνουν τα οικονομικά τους, αν ποσοτικοποιείται αν αυτά τα στοιχεία. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό ο κύριος Ρέν και ο κύριος Βράντεμάχερ γνωρίζει τις ενέργειες της λεγόμενης χρηματοοικονομικής μηχανικής για την τιτλοποίηση κάποιων στοιχείων από τα κράτη-μέλη που θέλουν κάπως να ψημιθιάσουν τους λογαριασμούς τους και να καλύψουν τα ελλείμματά τους μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Θα ήθελα λοιπόν αν αυτό το θέμα σας έχει απασχολήσει. Ποιες είναι οι ενέργειες τιτλοποίησης που γίνονται, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται και σε ποιο βαθμό τροποποιούν τα επίσημα στοιχεία για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος των χωρών της ζώνης του ευρώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ρέν, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδος η Κομισιόν έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας σας. Ως θεματοφύλακας των συνθήκων δεν είχε τη δύναμη παρά τις προειδοποίησεις της Eurostat να κάνει μια πλήρη εξέταση και έρευνας και επίσης δεν κατάφερε να συμφωνήσει για μια γρήγορη απόφαση στα θέματα αυτά. Έχουμε χάσει λοιπόν πάρα πολύ χρόνο. Την τελευταία εβδομάδα η, Ευρω... η Ελλάδα έχει υποστεί χωρίς να υπάρχει λόγος υπερβολικά επιτόκια και αυτό θίγει όλη την Ευρώπη. Επομένως θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Μήπως καταρχήν είναι πολλές χώρες και η δική μου χώρα περιλαμβάνεται σε αυτό τον ε, υπολογισμό, μήπως υπάρχουν χώρες οι οποίες με σκιώδεις προϋπολογισμούς αποκρύπτουν ένα μέρος του χρέους τους. Δεύτερον, υπάρχει μια ομοιόμορφη μεταχείριση από την Κομισιόν όλων των κρατών μελών και ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τους ισολογισμούς τους. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου λοιπόν και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Εάν εμείς κοιτάξουμε αυτό το οποίο προβλέπεται να γίνει όπως στο μέλλον, όπως είπε και η προλαλήσασα, είναι μονάχα η αρχή. Μιλάμε για μια υποστήριξη η οποία θα καλύψει τα επόμενα τρία χρόνια. Το επόμενο ερώτημά μου είναι για ποιο συνολικό ποσό μιλάμε και πότε θεωρείται σε συγκεκριμένο επίπεδο ότι η Ελλάδα θα ζητήσει αυτή τη βοήθεια. Μέχρι στιγμή δεν την έχει ζητήσει αυτή τη βοήθεια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει σύντομα αυτό το πράγμα. Θα γίνει κάποια στιγμή. Ποια θα είναι λοιπόν η διαδικασία όταν η Ελλάδα ζητήσει αυτά τα χρήματα και με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει σε μόνιμο επίπεδο να αντιμετωπίσει και μετά να εξέλθει από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Γενική Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε για τις εργασίες σας. Ε, ξέρουμε ότι δεν κατήχατε αυτή τη θέση τα περασμένα έτη. Τώρα θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο εξή ερώτημα. Πώς θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση στη συζήτηση είναι το εξή. Δεν είναι ότι δεν ξέραμε τι έγινε και σα παραπέμπω στην εξαιρετική έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Ιανουαρίου 2010, ειδικά για την Ελλάδα, όπου βλέπουμε ότι είχαμε επαρκή στοιχεία για να έχουμε και γνώση των προβλημάτων. Το πρόβλημα ε, ε, είναι ότι δεν θα ε, αναδιαμορφώσουμε την Ευρώπη τώρα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως το ευρώ δεν έχουμε παρικείς ελεγκτικές αρμοδιότητες ε, των ε, στατιστικολόγων της Eurostat. Έχουμε ένα χαλαρό συντονισμό, ένα, μια ανεπαρκή συνεργασία των ομοτήμων. Ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της συνεργασίας. Κύριε Ολυρένα έχετε την ευκαιρία τώρα να επηρεάσετε την αναδιαμόρφωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Έχουμε μία ε, πασιφανώς ανεπαρκή πολιτική 2020, μα πότε επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει κεντρικό ρόλο και θα προάγει το ευρωπαϊκό συμφέρον και θα σταματήσει να παίζει με τα κράτη-μέλη. Και δεν ε, το καταλογίζω μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πότε θα σταματήσει να παίζει με το μέλλον του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Γνώσης γενικότερα. Um, Ευχαριστώ. Ας περάσουμε στις απαντάσεις. Έχω άλλους 11 βουλευτές ε, που έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, δεν ε, θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε στον προβλεπόμενο χρόνο και θα υποφεληθούμε από το ότι έχει ακυρωθεί το τρίτο τμήμα της σημερινής ακρόασης. Κύριε Λιρέν, Πρόεδρε. Είναι δύσκολες οι ερωτήσεις, ταυτόχρονα όμως είναι και πολύ σημαντικές. Θα αρχίζω με τα σχόλια και τις ερωτήσεις του κυρίου Μπούλμαν. Με ρώτησε πώς ε, με ε, κοινοτική δράση μπορούμε να αναχαιτήσουμε κερδοσκοπικές επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο διοργανώσαμε αυτήν την σημερινή σημαντική συζήτηση για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το οπλοστάσιό μας, τα εργαλεία μας, την ετοιμότητά μας για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις στη ζώνη ευρώ. Παρότι δεν έχει γίνει επίσημη συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων, παρόλα αυτά ο πρόεδρος Μπαρόσο και οι συνάδελφοί μου με έχουν υποστηρίξει και έχω ε, λάβει εντολή για να εισηγηθώ μέτρα στους συναδέλφους μου. Όταν υποβάλλω τις προτάσεις μου στους Υπουργούς ε, Οικονομικών, ευελπιστώ ότι ε, οι προτάσεις μου θα τύχουν εξίσου θετικής αποδοχής. Έχετε δίκιο όταν μιλάτε για τις πληρωμές για τις χώρες εκτός ζώνης ευρώ και ότι τα όσα ισχύουν εκεί επηρεάζουν και την κατάσταση μέσα στη ζώνη ευρώ. Μιλάμε για ένα μηχανισμό διευκόλυνση τη δημοσιονομική σταθερότητα μέσα στη ζώνη ευρώ που ε, βασίζεται στην ε, ε, αυστηρή αιρεσιμότητα, αυστηρούς κανόνες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης και για την λήψη της χρηματοοικονομικής αρρωγής. Δεν είχαμε συμφωνήσει τίποτα πριν την περασμένη Κυριακή. Τώρα έχουμε μία συμφωνία για να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη που προκύπτει άμεσα. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής ακρόασης εξάλλου, ότι χρειαζόμαστε καλύτερο εξοπλισμό, ε, καλύτερα εργαλεία για ενδεχόμενες μελλοντικές ε, κρίσεις. Και ξαναλέω, θα υποβάλω επίσημη συγκεκριμένη πρόταση για τον ε, μηχανισμό ε, στήριξης της δημοσιονομικής σταθερότητας μέσα στη ζώνη ευρώ. Δεύτερον, κυρία Ποδηματά και κύριε Αργάγιο, για τα swaps, για τις συμφωνίες ανταλλαγής και τα στατιστικά στοιχεία. Ε, θα το αφήσω το θέμα στο συνάδελφο τον Walter Rademacher γιατί γνωρίζει εις βάθος αυτό το ζήτημα διότι το έχει ερευνήσει εις βάθος. Θα πω μόνο ε, με την ε, ιδιότητα του αρμοδίου επιτρόπου αρμοδίου για τη Eurostat δηλαδή, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα ζητήσω από τη Eurostat και από το Βάλτερ να εργαστούν και παρά τις νέες πληροφορίε που θα πάρουμε από την Ελλάδα, καθημερινά εξάλλου λαμβάνουμε νέες πληροφορίε από την Ελλάδα, αλλά δεν γίνεται εβδομαδιαίως ή καθημερινά αναθεώρηση των ε, στοιχείων λόγω της ευαισθησίας ε, της ε, κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί στις αγορές για την έκδοση χρέους και για τα swap στις συμφωνίες ανταλλαγής θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση μία και έξω και θα δούμε πώς επηρεάζει το χρέος. Γιατί ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν επηρεάζει το επίπεδο του χρέους σήμερα. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και οι ελληνικές αρχές, ξαναλέω, έχουν βελτιώσει σημαντικά ε, τον τρόπο εργασίας τους. Ε, θα το επιβεβαιώσει, φαντάζομαι, ο Βάλτερ, αλλά έχουμε επαρκή δεδομένα πιστεύουμε ε, για το έλλειμμα και έχουμε και συγκρίσιμα αξιόπιστα δεδομένα σε σχέση δηλαδή με το χρέος ε, άλλων χωρών. Για τις ερωτήσεις ε, του κυρίου Κλίντς και της κυρίας Ποδήματα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν την Κυριακή δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για να σας εξηγήσω λεπτομερώς τι έγινε. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση και το τονίζω ότι χρειαζόμαστε γιατί πρέπει να πείσουμε τις αγορές ότι έχουμε έναν ε, ξεκάθαρο σαφή μηχανισμό που θα δώσει στήριξη αν χρειαστεί. Τώρα διαπραγματευόμαστε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αρχίσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη και θα συνεχίσουμε τις προσεχείς ε, ημέρες ε, για τα ε, προγράμματα εκταμίευσης με δόσεις, το υπονομεζόμενο conditionality. Λοιπόν, την Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην συνεργασία με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο θα αποτιμήσουν τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα ε, για να ενεργοποιήσουν ενδεχομένως ε, τον ε, μηχανισμό και θα υπάρχει εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διαπραγματευτεί συμφωνία δάνειοδοσίας και θα συντονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα διμερεί δάνεια εάν ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από το Eurogroup ε, φυσικά. Πάντως ε, έχει προσδιοριστεί σαφώς ε, ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια αυτής της εντολής γιατί πλέον έχουμε σαφή εντολή. Και τώρα επανέρχομαι σε κάτι που ανέφερε ο κύριος Μπούλμαν Εφόσον δεν υπάρχει κοινοτικό όργανο, αποφασίζουν ε, τα κράτη-μέλη. Και έτσι απαντώ και στον κύριο Κλίντ. Μέσα σε δύο-τρει μήνε ε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση, με δυσκολία ομολογουμένω. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά Και ξέρετε ότι η πολιτική δείχνει, είναι η τέχνη του ε, δυνατού ε, και αυτό φάνηκε γιατί καταφέραμε να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Ποιο είναι το πακέτο. Η συμφωνία προβλέπει ότι δεσμεύονται τα κράτη-μέλη ε, της Ευρωζώνης για 30 δις τον πρώτο χρόνο ρήξη θα υπάρξει συναπόφαση και συγχρηματοδότηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που φυσικά είναι αυτοδύναμο για το ποσό που θα διαθέσει το ίδιο. Και για το δεύτερο και τρίτο έτος αυτού του τριετού σε προγραμματος προγράμματος 2011-2012 ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤΕ και το Διεθνέ Ενομισματικό Ταμείο θα συνεργαστούν φυσικά με την ελληνική κυβέρνηση για την αναχρηματοδότηση του δανείου σε περίπτωση ξαναλέω που θα χρειαστεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού. Κυρία Γκουλάρτ, είπατε πώ δεν έχει αναλάβει δράση η Επιτροπή για την Ελλάδα. Μάλλον απλουστεύω αυτά που είπατε. Δεν το νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δείτε τις δύο βασικές διαστάσεις, δηλαδή δημοσιονομική εξυγίανση στην Ελλάδα φαινός και αφετέρου δημοσιονομική αρρωγή αν χρειαστεί. Μα έχουν δρομολογηθεί, δρομολογηθεί και τα δύο. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν έχει αναλυφθεί δράση. Φυσικά δεν έχουμε επιτύχει τον τελικό στόχο. Υπολείπεται μεγάλο έργο και για την ελληνική κυβέρνηση και για το ελληνικό κοινοβούλιο και για τη δημόσια διοίκηση καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Πάντως, ξαναλέμε, έχει δρομολογηθεί για φέτος η δημοσιονομική εξυγίανση. Θα ε, έπονται και άλλα μέτρα το 2011 και 2012, αλλά έχει κινηθεί διαδικασία. Και δεύτερον, για το μηχανισμό... Ε, χρηματοοικονομικής υποστήριξης ε, θέλουμε η, πρόταση να μετατραπεί σε έναν πιο πάγιο, πιο μόνιμο μηχανισμό αρρωγής. Ε, μιλήσατε για το δικαίωμα πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, μη χρήση του δικαιώματος, ε, πρωτο, μη άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας. Στους Financial Times πριν από λίγες μέρες ένας αξιωματούχος κράτους μέλους που δεν αναφέρεται ονομαστικά, εγώ υποψιάζομαι ποιος είναι τέλος πάντων, είπε τα εξής. Τα κράτη-μέλη είναι ε, οι δεσπότες, αν θέλετε, της συνθήκης ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο υπηρέτης. Δεν έχω πρόβλημα να είμαι υπηρέτης ε, σεβαστό το επάγγελμα. Εμεί είμαστε θεματοφύλακες ε, τη συνθήκη και φυσικά έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλία και πιστέψτε μας ε, θα το ασκήσουμε. Um, yes, maybe I come uh, to the of uh, of uh, Να έρθω συγκεκριμένα στο θέμα των ε, ισοζυγίων και το ποιοι ήταν οι κανόνες των ισολογισμών, συγγνώμη. και το ποιοι είναι οι κανόνες αλλά και πώς εξελίχθηκαν αυτοί. Σημείο κίνηση να σας πω ότι στον τομέα μας υπάρχει ε, αλληλεπίδραση ανάμεσα στην θέσπιση κανόνων και τη νέα συμπεριφορά. Τα νέα δηλαδή δημιουργικά μέσα και η αντίδρασή τους σε σχέση με τους κανόνες. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν και στην αρχή αυτής της δεκαετίας και θα είναι φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύσει μάλλον και για τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή, οι εξελίξεις δεν θα σταματήσουν και εμείς ως στατιστικολόγοι είμαστε πάντοτε πίσω από τις εξελίξεις κατά κάποιο τρόπο και να προσπαθούμε δηλαδή να καλύψουμε τα νέα μέσα δημιουργώντας νέους κανόνες. Τούτου λεχθέντος βέβαια, σε δύο επίπεδα υπάρχουν οι γενικοί κανόνες οι οποίοι ορίζονται από τους κανονισμούς και ο κανονισμός εδώ άλλαξε το 2000 αλλά η αλλαγή αυτού του κανονισμού δεν κάλυπτε δεν αγκάλιαζε ολόκληρη την αγορά των swaps. Έχουμε έναν γενικό κανονισμό για τα swaps, αλλά όχι το φαινόμενο των συνθήκων εκτός αγοράς. Αυτό πήρε κάποιο χρόνο. Και το 2008, σε δεύτερο επίπεδο, όπου έχουμε δηλαδή τι κατευθυντήριε γραμμέ, καθώ και ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι συμπεφωνημένο μεταξύ κρατών μελών τη Eurostat και μετά ε, δημοσιεύεται και από την Eurostat. Οι κανόνες λοιπόν άλλαξαν. Μετά από το 2008, η καταγραφή των swap εκτός αγοράς ε, είχε σαφώς καθοριστεί και έκτοτε είναι σαφές πως και η συμπεριφορά των ε, ε, χωρών άλλαξε γιατί δεν υπήρχαν τα ίδια κίνητρα. Άρα λοιπόν οι χώρες τα κατέγραφαν όλα αυτά αντιστοίχω. Μετά όμως από την αλλαγή των κανόνων, ρητά ζητήσαμε και από τα 27 κράτη-μέλη να μας αναφέρουν εάν κάνουν τέτοιου είδου επιχειρήσει ή όχι, συναλλαγέ ή όχι. Και στην ελληνική περίπτωση έχουμε μια επιστολή με σφραγίδα που έλεγε ότι αυτού του είδου οι συναλλαγέ δεν είναι νόμιμε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Άρα λοιπόν εκεί δεν μπορούσαμε να ψάξουμε περισσότερο γιατί δεν είχαμε τις κατάλληλες αρμοδιότητες. Σε εκείνη τη φάση απλά έπρεπε να πιστέψουμε αυτό που μας είπαν. Ένα σύντομο ερώτημα. Ρώτησα αν υπήρχαν άλλα κράτη-μέλη που χρησιμοποίησαν αυτές τις ε, ενέργειες και αν ξέχετε στοιχεία που δείχνουν ότι στις συναλλαγές αυτές είναι πλάκι η Goldman Sachs. Υπήρξαν άλλα κράτη-μέλη ή, ή κράτη-μέλη που έκαναν ανακοίνωση στην Κομισιόν για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ερώτημά σας. Τώρα, το ερώτημα, ε, ποιες τράπεζες θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω μία απάντηση. Ζητώ την κατανόησή σας. Αλλά η, είναι πολύ πιθανό ότι δεν πρόκειται μονάχα για την Goldman Sachs, κατά πάσα πιθανότητα. Και ναι, πράγματι υπήρξαν και άλλες χώρες οι οποίες έκαναν τέτοιου είδους ενέργειες Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο και Γερμανία. Είναι οι χώρες οι οποίες έκαναν τέτοιες ενέργειες και φυσικά και η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια υπόθεση που είναι μια περίπτωση που ακόμα πρέπει να την διευκρινίσουμε πλήρω, για να το πω καλύτερα. Θα τα πω πάλι στα αγγλικά. Έχουμε μετάφραση. Να επαναλάβω την απάντησή μου στα αγγλικά. Όχι, την ακούσαμε στα αγγλικά. Όχι, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε και δεν έχουμε και χρόνο. Θα συνεχίσετε να απαντάτε στις υπόλοιπες ερωτήσεις που έθεσαν ε, ο κύριος Γκαρσία Μαργκάλη, που είπε ότι ήθελε κάποιες λεπτομέρειες για τα ομόλογα. Ναι. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, κύριε Διευθυντά. Γνωρίζει η Eurostat ότι υπήρξαν ενέργειες τίτλοποίησης σε κάποιο κράτος μέλος που επηρεάζουν τα στοιχεία του δημόσιου χρέους, του, του, του ελλείμματος μάλλον που έχουμε υπόψη μας ή όχι. Ναι, γνωρίζουμε για την τιτλοποίηση υπάρχει μια ε, κατευθυντήρια γραμμή, μια και αφού εκδόθηκε αυτή δεν δήλωσε κανένα κράτος μέλος ότι χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ε, μηχανισμό, τιτλοποίηση δηλαδή. Με, πριν από την έκδοση της συγκεκριμένης κατευθύνης γραμμής υπήρχε ε, γινόταν τιτλοποίηση. Αυτή τη στιγμή, μετά την έκδοση αυτή ε, τη κατευθύνια γραμμή, δεν έχουμε δήλωση από κανένα κράτο που να λέει ότι προχωρεί σε τιτλοποίηση. Έχουμε φυσικά την παράταση των περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί θα μπορούσε να στείλει ο Γενικό Διευθυντή τη Eurostat στην Επιτροπή μα και στο Κοινοβούλιο ένα πλήρη κατάλογο των ενεργειών τιτλοποίηση που έχουν γίνει στο παρελθόν από, ένα, από κάθε ένα κράτο μέλο. Okay. Μάλιστα. Όταν αφορά τις ε, εκτός ισολογισμού ή κρυφές ε, συναλλαγές, και την καταγραφή του χρέους, Έχουμε φτιάξει ένα πακέτο που ασχολείται με τα φαινόμενα της, ε, δημοσιονομικής, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο εύρος διαφόρων συναλλαγών και είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνουμε ανάμεσα στις ε, ενδεχόμενες, ε, στις ενδεχόμενες ζημιές και τις πραγματικές ζημιές. Και για να διασφαλίσουμε 100% διαφάνεια για όλους τους χρήστες των στατιστικών μας, έχουμε επεκτείνει τις ε, εκθέσεις στοιχείων με, έναν, με επιπλέον πίνακα που επιτρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα κάθε είδους ε, γενικών εγγυήσεων που μπορεί να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη. Αλλά Όλα αυτά τα προγράμματα εγγύησεων δεν έχουν οδηγήσει στην καταγραφή του χρέους ε, απαραίτητο. Ορισμένα από αυτά περιμένουν ε, για να καταγραφούν ε, είτε στο έλλειμμα είτε στα αντίστοιχα, στις αντίστοιχες στήλες καταγραφής του χρέους. Σας προτείνω λοιπόν να διαβάσετε αυτό το πίνακα διότι είναι πολύ φιλόδοξος και διαφωτιστικός. Uh, Ωραία, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως έχουμε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Γι' αυτό και θα ακούσουμε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Παρακαλώ να μείνετε στο ένα λεπτό. Γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβουν όλοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις. Δεν σας επιτρέψω να καταπατήσετε το χρόνο των συναδέλφων. Uh, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Επιτρέψτε μου... Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω κάτι στο σώμα. Πριν από δύο μήνες, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, σε σχετική ερώτηση για τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδος, και αυτό που θα πω δεν νομιμοποιεί καθόλου την Ελλάδα, για οτιδήποτε έκανε με τα στατιστικά της στοιχεία, το διευκρινίζω. Σε σχετική ερώτηση λοιπόν προς τον πρόεδρο Μπαρόσο, γιατί δεν έδωσε δικαιοδοσία λογιστικού ελέγχου στην ε, Eurostat, είπε ότι το ζήτησε, απήντησε ο πρόεδρος ως εξής. Το 2004 ζήτησε από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωζώνης να επεκταθεί η λογιστική δικαιοδοσία στη Eurostat και η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων αρνήθηκε τον λογιστικό έλεγχο, την ε, δικαιοδοσία λογιστικού ελέγχου από τη Eurostat. Βλέπω, κυρία Πρόεδρε, ότι σιγά σιγά ανοίγει ένα κουτί της Πανδώρας εδώ σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Επίτροπε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Εδώ πλέον μετά από τους τρεις μήνες δεν συζητάμε για το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, αλλά ε, συζητάμε για κίνδυνο στην Ευρωζώνη. Αν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα αυτών που αποφασίσατε την Κυριακή, θα μας διευκόλυνε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ερώτησή μου απευθύνεται στον Επίτροπο κύριο Ρέν ε, και θα είναι πολύ σύντομη. Παρακαλώ να μας πείτε εάν σε περίπτωση ενεργοποίησης του Μηχανισμού Οικονομικής Στήριξης για την Ελλάδα η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προηγηθεί της χρηματοδότησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή το αντίθετο. Ευχαριστώ. Μιλάμε για τις ε, συμφωνίες ανταλλαγής και την τιτλοποίηση. Το ερώτημα όμως είναι πιο βασικό. Γνωρίζει η Κομισιόν ότι υπάρχει ένα μέλος της Ευρωζώνης του οποίου η κυβέρνηση και το σύστημα ε, λογιστικής βασίζεται σε μια λογιστική ταμιακών ροών και όχι καταβεβλημένων. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μέρος, μέλος της Ευρωζώνης και το οποίο μπορεί κανείς να χειραγωγήσει το έλλειμμα διότι η κυβέρνηση μπορεί να περιμείνει για την καταβολή κάποιων πληρωμών οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και καταβληθεί. Ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος στη σειρά, κύριε Χουντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω την εντύπωση πως η, η αξία αυτής της δημόσιας ακρόασης αρχίζει να φαίνεται στην εξέλιξη που αρχίζουμε από τα εύστοχα ερωτήματα των συναδέλφων να παίρνουμε κάποιες απαντήσεις. Η δική μου η ερώτηση έχει το εξής σκεπτικό. Η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε αναξιόπιστη διότι επί χρόνια αλλίωνε τα στατιστικά δεδομένα και διότι χρησιμοποιούσε, αν αυτό είναι ο σωστός μεταφραστικός όρος, χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να αλλοιώνει την εικόνα του χρέους. Για αυτή τη συμπεριφορά τιμωρείται σήμερα, ανάμεσα σε άλλους λόγους ενδεχομένω, με δυσκολίες δανεισμού και υψηλά σπρέτζ. Το ερώτημα που προκύπτει και από τις απαντήσεις που λήφθησαν, τι γνώριζαν οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Κομισιόν και της Eurostat για τις λογιστικές αλχημίες που έκανε η Ελλάδα για αυτές τις μορφές αλλίωσης του δημόσιου χρέους που έκανε η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες όπως φάνηκε από την απάντηση που μας δόθηκε. Υπάρχουν ευθύνε των πολιτικών προϊσταμένων. Εδώ υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δια παραλήψεων ή διαπράξεων συνέπραταν συνειδητά στην αλλίωση αυτών των στοιχείων. Η Μοντ στις 2 Μαρτίου μιλάει για πρώην επιτρόπους και πρώην στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα έχουν στελεχική ιδιότητα στην Goldman Sachs. Κατόπιν τούτου το ερώτημα είναι προβλέπετε κάποια διαδικασία απόδοσης ευθυνών αυτών των πολιτικών προϊσταμένων που γνώριζαν, μετήχαν ή δεν μετήχαν στην αλλίωση αυτών των δεδομένων. Και το δεύτερο ερώτημα. Η Ελληνική Βουλή συζητάει να φτιάξει μια εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει αυτό το θέμα. Αν κληθούν αυτοί οι πολιτικοί προϊστάμενοι, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τι γνώριζαν και τι δεν γνώριζαν για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ. Hans Peter Martin. Hans Peter Martin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε σαν πεπισμένος υποστηρικτής του Ευρώπου ανησυχεί, θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Κύριε Ρεν, κατάλαβα καλά την απάντησή σας για τον Βολφ Κλίντς, που ότι επιβεβαιώνεται αυτά που λέει το Handelsblatt, ότι η χρηματοδότηση δεν θα είναι 30 μονάχα δισεκατομμύρια, αλλά συνολικά 90 δισεκατομμύρια η Κομισιόν έχει ήδη πάρει μια απόφαση για το 2011 και το 2012. Εάν υπάρξουν λοιπόν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα είναι με την ίδια ποσόστοση 8,4 δισεκατομμύρια παραγωγικά το χρόνο για τη Γερμανία και αντίστοιχα για τις άλλες χώρες. Είναι ορθά αυτά. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει καλύψει επομένως τα επόμενα τρία χρόνια. δεύτερο για τον κύριο Ράντε Μάχα έχετε την συμπαράστασή μου γιατί βρισκόσαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το θέμα αυτό των συμφωνιών ανταλλαγής, των swaps. Πώς έχετε αντιδράσει όταν αναλάβατε τα, όταν μάθατε για αυτά τα στοιχεία και πώς αντιδράσατε ενάντια των πολιτικών υπευθύνων της Επιτροπής. Μας τελειώνει ο χρόνος, λέει η Πρόεδρος θα δεχτώ ερωτήματα, αλλά αν δεν βιαστείτε δεν θα μπορέσουν να υπάρχουν να απαντήσει. Κυρία Φερέιρα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εγώ θέλω να θέσω την εξή ερώτηση. Σήμερα, στο τέλο τη ε, συνέντευξη τύπου, ε, το Associated Press έθεσε ω μεγάλο πρώτο σημείο, ω ε, τίτλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει η Πορτογαλία να προετοιμαστεί για περαιτέρω περικοπέ στον προπολογισμό. Το πρόγραμμα σταθερότητα τη Πορτογαλία παρουσιάστηκε. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα όπου δεν υπάρχουν κανένα είδους απάτες, ε, τουλάχιστον γνωστές μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μέχρι το 2005 και το 2007 το έλλειμμά μας ε, περιορίστηκε στο 2,5. Φαίνεται να είναι υποδειγματική η συμπεριφορά μας. Δεν θεωρεί η Κομισιόν ότι ήταν καλύτερο, προτιμότερο να πούμε ναι, εμείς δεχόμαστε αυτά που προτείνει η χώρα και εμπιστευόμαστε τη χώρα πως ε, θα κάνει κάποια μεταρρύθμιση με την ε, αγορά που είναι τόσο ευαίσθητη αυτή τη στιγμή με τους ε, κερδοσκόπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν με τα... το χρέος κάθε χώρας. Ε, δεν νομίζετε πως μια τέτοια δήλωση δεν είναι και πολύ σωστή. Δεν είναι αυτό ένα από τα διδάγματα που αποκομίσατε από την ελληνική εμπειρία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να μου εξηγήσετε και ποια είναι η θέση σε σχέση με την Πορτογαλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά από τα ερωτήματα που είχα στο μυαλό μου έχουν ήδη απαντηθεί, αλλά θα ήθελα να εστιάσω στο γεγονός ότι μετά από την Ένρον οι όμιλοι υποτίθεται ότι θα τροποποιούσαν τη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, ακούμε πως η τιτλοποίηση γίνεται, εξακολουθεί να γίνεται από τα κράτη-μέλη μας συμπεριλαμβανωμένων των διαφόρων ε, των, ε, των χρημάτων, διαφόρων ε, λαχείων, και φαίνεται πως βρίσκουν διάφορους μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης ε, είτε με ειδικά οχήματα. Ένα σωρό ακροστοιχίες φαίνεται να χρησιμοποιούνται όλη την ώρα. Δεν υπάρχει ένα μορατόριο για τα κράτη-μέλη ώστε να επανυποβάλλουν τα στοιχεία τους με ένα ξεκάθαρο τρόπο ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα επίπεδα χρέους του καθενός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πράγματι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Έπινγκ, του συναδέλφου μου, για το συγκεκριμένο αυτό το θέμα που έθεσε, που το έθεσε και η Επίτροπος, η Καγκελάριος Μάλλον για το αν πρέπει να αναπτυχθεί μια νομική διαδικασία, ώστε μια χώρα η οποία κατά συρροή και κατά επανάληψη ε, παραβιάζει τους κανόνες, θα αναγκαστεί να φύγει από τη ζώνη του ευρώ. Για το θέμα τώρα των ποινών θα ήθελα να υπάρξει υποστήριξη από τους για τις χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με τα διαφθορτικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από ό,τι γνωρίζω 18 δισεκατομμύρια ευρώ ποσά για διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί, τα οποία μπορούν να πληρωθούν στην, Ευρώπη, στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Η Κομισιόν θα μπορούσε να απαιτήσει να μην πληρωθούν τα ποσά αυτά, να εμποδίσει να πληρωθούν τα ποσά αυτά σε μια χώρα η οποία παραβιάζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά υπάρχουν και φήμες στον τύπο ότι μπορεί κανείς να φανταστεί μια διαδικασία ταχεία οδού για να υπάρξει μια αποδυνάμωση της διαδικασίας συμμόρφωσης ώστε να εκταμιευτούν τα λεφτά αυτά ταχύτερα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα θέματα. Δύο σύντομα ερωτήματα λέει ο κύριος Λάγκεν προς τον κύριο Επίτροπο. Καταρχήν μετά από αυτό που ζήτησε να μάθει ο κύριος Κλίντς συζητούμε εδώ και πολύ καιρό για τις αιτίε και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα του συστήματος ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πώς θα το εξασφαλίσουμε και θα το κάνουμε πιο εύρωστο. Ποιες είναι οι προτάσεις της Κομισιόν. Και εδώ βλέπω να υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Όταν ο κύριος ε, Ρεν είπε για την Πορτογαλία ότι χρειάζονται οπωσδήποτε περαιτέρω εξηγιάνσει στο επίπεδο του προπολογισμού, αλλά ήδη από την άλλη πλευρά λέει ότι η Πορτογαλία είναι αξιέπαινη διότι έχει συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα με 740 εκατομμύρια ευρώ. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ έχουμε και τον εκπρόσωπο της Goldman Sachs, ο οποίος θα λάβει το λόγο στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν είναι πράγματι γνωστό σε εσά ότι ορισμένοι θέλουν να κάνουν ε, αγωγή κατά της ε, Goldman Sachs για τον τρόπο με τον οποίο τιτλοποίησε στοιχεία κρατικού χρέους. Και αυτό αφορά φυσικά και την Ελλάδα. Ο Όλι Σμιτ, ευχαριστώ. Σε σχέση με το παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, ίσως εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε ως κοινοβούλιο ότι και εμείς έχουμε κάποια ευθύνη στα θέματα αυτά. Ορισμένοι από εμά ε, στην ουσία ψηφίζαμε και δεχτήκαμε την Ελλάδα να μπει στην Ευρωζώνη. Ίσως λοιπόν και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια ευθύνη. Με τα πω τώρα σου ειδικά. Γιατί ξέρω πως ο Επίτροπος Ρεν μιλά πολύ καλά τη γλώσσα αυτή. Θέλω να ξέρω τι γίνεται με τους μηχανισμούς αυτούς, που, αυτό, μηχανισμό μάλλον αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Φαίνεται εξαιρετικά εφισ η Κομισιόν έχει λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις χώρες που είναι εκτός του ευρώ. Και να δούμε ποια είναι η δική τους κατάσταση. Πώς αυτές θίγονται από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωζώνη γιατί υπάρχει αντίκτυπος στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Στη χώρα μου επίσης συζητάμε για την περίπτωση της Ελλάδας και ο Επίτροπος Ρεν δεν πιστεύει πως θα ήταν λογικό να συμμετέχουν και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης στα δάνεια και στις εγγυήσεις και αυτό σε ένδειξη ελεγγύης μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Πρόεδρος. Κι άλλοι μου ζητούν το λόγο, δεν σταματάτε, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να πάψουμε πια με τις ερωτήσεις για να μπορέσει ο Επίτροπος να απαντήσει. Θα έρθει και στην επόμενη μας συνεδρίαση, θα μείνει μάλλον και στην επόμενη μας στην υπόλοιπη συνεδρίαση και ίσως θα μπορούσε στη συνέχεια να απαντήσει. Είπατε ότι θα βασιστείτε στο άρθρο 136 της συνθήκης, ενώ το Κοινοβούλιο θα ήθελε να προχωρήσετε με πιο γενικό τρόπο και να χρησιμοποιήσετε το 121, όπου θα εμπλακεί και το Κοινοβούλιο στην πόλημερη εποπτεία. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε ίσως να βρει σύμφωνο τον κύριο Σμιτ με βάση αυτά που, ρώτησε, που ζήτησε. Ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Τζαβέλα. Σε σχέση με τις ελληνικές στατιστικές και την ερώτηση που έθεσε το Κοινοβούλιο στον κύριο Μπαρόσο. Εγώ μπορώ μόνο να αναφερθώ στο γεγονός ότι την τελευταία φορά τα κράτη-μέλη δεν ήταν έτοιμα να δώσουν στην Επιτροπή τις κατάλληλες αρμοδιότητες. Φαντάζομαι πως και τα κράτη-μέλη έχουν αποκομίσει τα δάγματα της κρίσης και πως αυτή τη φορά θα δώσουν τις κατάλληλες αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να ενεργήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο θα μπορεί να λάβει τη σχετική απόφαση οποτεδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή είναι μια πολύ ε, Συμπαγή και στέρεα πρόταση έχει ήδη συζητηθεί πριν από πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ουσιαστικό λόγος να μην υιοθετηθεί πολύ σύντομα. Σε σχέση τώρα με το χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διακυβέρνηση στην οποία αναφερθήκατε, τουλάχιστον στα αγγλικά αυτό άκουσα, ότι περιμένουμε τρεις μήνες, μα 30 χρόνια περιμένουμε διότι το θέμα αυτό έχει ήδη θυγεί σε πάρα πολλές εκθέσεις, ε, για να σας αναφέρω μόνο μία, την έκθεση Delors που μετά οδήγησε στην Νομισματική Ένωση. Αυτά αυτές οι προκλήσεις είχαν εντοπιστεί από τότε. Τώρα έχουμε μάθει τα διδάγματα βέβαια, δεχτήκαμε πολύ γερά χτυπήματα, αλλά Γι' αυτό και μιλάμε για το μηχανισμό επίλυση ε, αντιμετώπιση κρίσης αλλά και την σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδου μηχανισμού στη διάθεσή μα για να δυσφαλίσουμε την σταθερότητα στην Ευρωζώνη υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ωστόσο ταυτόχρονα χωρί να μπω τώρα στην επίρρηψη ευθυνών ε, να μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα ζει εδώ και χρόνια, έζουσε ε, μάλλον εδώ και χρόνια πάνω από τα, τις δυνατότητές της. Και υπήρξαν πολλές αντικανονικότητες εδώ και χρόνια. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Τώρα, Κοιτάξτε τώρα, για την ε, έκτη και το δούνο του δεν έχει κάνει ακόμα αίτηση η ελληνική κυβέρνηση, οπότε δεν ξέρουμε ποια θα είναι ε, το αίτημα. Πάντως υπάρχουν ε, οι όροι, έχουν ήδη συμφωνηθεί. Ακόμα δεν έχει ζητηθεί όμως αυτή η βοήθεια. Ο κύριος Κικόνα αναφέρθηκε σε μια χώρα η οποία χρησιμοποιούσε παλαιομοδίτικες τρόπους ε, λογιστικής και τα λοιπά και Ίσως ο κύριος Ρόντεμα έχει να αναφερθεί σε αυτή τη χώρα. Εγώ ζήτησα και εγώ ίδιος πληροφορίες από την Eurostat. Έπειτα αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η Ελλάδα τιμωρείται. Εγώ δεν το βλέπω με τέτοιο τρόπο και η απόφαση της περασμένης ε, Κυριακής είναι έκφραση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Υπήρξε και το ερώτημα του αν υπήρξαν πλημελείς ενέργειες ε, και κατά πόσο υπάρχουν ε, εξεταστικές επιτροπές για να δούμε ποιες ήταν οι στατιστικές ε, ενέργειες, πράξεις και η αλλίωση στοιχείων. Εγώ έχω ζητήσει τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής και η απάντηση μέχρι στιγμής ήταν όχι, γιατί τότε που γίνονταν ήταν νόμιμες οι ενέργειες αυτές. Μπορεί να μην φαίνονται και τόσο θεμητές αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν νόμιμες σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους. Και τώρα από το 2008 και έπειτα η Eurostat καταγράφει όλο αυτού, αυτές του είδους τις ενέργειες. Το 2008 άλλαξαν τα πράγματα, διορθώθηκε η κατάσταση, αλλά θεμητό δεν σημαίνει νόμιμο. Επίσης, ρώτησα όλους τους διευθυντές μου να δω κατά πόσο σε οποιαδήποτε αποστολή έχουν διαπιστώσει παρανομίες ή πλημελείς ενέργειες. Αυτό πρέπει να γίνεται άμεση ενημέρωση δική μου, αλλά δεν έχει γίνει. Ο κύριος Μάρτιν αναφέρθηκε σε κερδοσκοπία. Σε εικασίες κερδοσκοπίας δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεν υπάρχει βάση. Να πω μόνο πως Εάν ο μηχανισμός οικονομικής συναρρογή προς την Ελλάδα δεν ενεργοποιηθεί, είναι σαφές πως τον πρώτο χρόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν δεσμευθεί μέχρι 30 δις ευρώ. Ταυτόχρονα ε, θα υπάρχει χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα ποσά τώρα θα τα αποφασίσει μόνο του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έπειτα για τα δεύτερο και τρίτο έτος αυτού του πολιετούς, του τριετούς προγράμματος, πιθανές αποφάσεις ε, θα λαμβάνονται επί τη βάση της αξιολόγησης που θα κάνει η Κομισιόν και η ΕΚΤ προς την ε, Υπουργούς Οικονομικών του Ευρωγκρουπ. Ερώτηση για την Πορτογαλία από την κυρία Φέρειρα. Σήμερα εξετάσαμε το πρόγραμμα σταθερότητας της Πορτογαλίας που έφτασε αργά και είμαι ευγνώμων στους υπαλλήλους μου που βοήθησαν ώστε να το μελετήσουμε, εργάστηκαν νυχθημερών. Σεβόμαστε τους κανόνες, ε, θέτουμε σε εφαρμογή τα όσα διακηρύττουμε και είναι σημαντικό κάθε πρόγραμμα σταθερότητας να αξιολογείται σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη, και αυτό κάναμε. Και όλα θεωρούμε πως η Πορτογαλική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο και πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σταθερότητας προς την οικονομική παγίωση περιλαμβάνονται κάποιοι κίνδυνοι όσον αφορά τα στοιχεία του 2009, όσον αφορά το έλλειμμα του δημόσιου τομέα και όσον αφορά την συνεχιζόμενες μακροοικονομικές εξελίξεις. Εάν υπάρξουν κίνδυνοι σε σχέση με τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ε, εξελίξεις, τότε ίσως να χρειαστεί προσαρμογή για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος σταθερότητας της Πορτογαλίας. Η κυρία Φόρτα αναφέρθηκε στην ερώτηση του κυρίου Έπινγκ για το αν μια ε, χώρα η οποία κατά συρροή και κατά επανάληψη ε, παραβιάζει το σύμφωνο σταθερότητας μπορεί να βγει από την Ευρωζώνη. Να αναφερθώ σε αυτά που γνωρίζω για τις συνθήκες, κανονικά αυτό απαιτεί αλλαγή της συνθήκης. Και όλοι γνωρίζουμε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Εγώ προτείνω, θεωρώ ότι ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων θα βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες αυστηρές προβλέψεις, ώστε να είναι τόσο λίγο ελκυστικός που καμιά χώρα να μην θέλει να το χρησιμοποιήσει. Εγώ θα πρέπει να σας πω προσωπικά πως έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την επιλογή καναγκαστικής εξόδου, γιατί αυτό δεν είναι σύμφωνα με τη συνθήκη. Εξάλλου, η φιλοσοφία των ιδρυτών πατέρων της Ένωσης δεν ήταν αυτή. Δεν συμφωνεί δηλαδή, δεν συνάδουν όλα αυτά. Ε, μάλλον κάτι τέτοιο με την αρχική φιλοσοφία. Ο κύριος Λάγκη ρώτησε πότε θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες Ήθελα να συζητήσω με το Κοινοβούλιο, ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχα. Θέλω να το συζητήσω και με το Συμβούλιο και θέλω επίσης να διαβουλευθώ με τους ενδιαφερόμενους φορείς από αυτού και σε λίγες εβδομάδες θα προβούμε σε ουσιαστική και συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να διευρυνθεί οικονομική εποπτεία και να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης των κρίσεων. Για την Πορτογαλία, στην οποία αναφερθήκατε ήδη απάντησα και το θέμα είναι κατά πόσο θα χρειαστεί να ληφθούν ε, ε, ε, επιπλέον μέτρα εάν προκύψει ο κίνδυνος, αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Επίσης να πω ότι η επίρρηψη ευθυνών δεν είναι πολύ παραγωγικός τρόπος για την ανέβρεση λύσεων και όσον αφορά το κατά πόσο η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο την Ευρωζώνη, η απάντησή μου είναι φυσικά θα πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια ένωση 27 κρατών μελών και οφείλουμε αυτό να θεωρούμε ως σημείο εκκίνησης. Αναφερθήκατε και η κυρία Πρόεδρος αναφέρθηκε 121, στο άρθρο 121 που είναι η προτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Συμφωνώ πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 121 όσον αφορά για παράδειγμα <coughs> τις οικομευρίες οικονομικές κατευθύνες γραμμές, τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, την ε, πιο αυστηρή στις πιο αυστηρές ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, την πρώιμη προειδοποίηση, την έγκαιρη μάλλον προειδοποίηση. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο αρκετά στο παρελθόν. Είναι ένα από τα μέσα λοιπόν που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο και αυτό αφορά και τα 27 κράτη-μέλη. Τούτου λεχθέντο, ε, εργαζόμαστε επί τη βάση τη συνθήκη Η συνθήκη είναι σαφή. άρθρο 136 καλύπτει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνη. Και εγώ θέλω να καλέσω τι χώρες που ανταποκρίνονται στις όρου για να γίνουν μέλη της Ευρωζώνη να το πράξουν, ώστε να είναι μέλη της ενισχυμένης ε, διακυβέρνησης. Να σας ρωτήσω αν στις τελευταίες σας απαντήσεις είπατε ότι έχετε ζητήσει από τα 27 κρατη να αναφέρουν τις συναλλαγές τους. Αυτό καλύπτει το είδος του μορατόριου που αναφέρθηκε όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, ισολογισμού. Ε, εκτός ισολογισμού, συγγνώμη. σω ο κύριο Ρόντε Μάκερ να μπορούσε να απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Ναι, ο κύριο Ρόντε Μάκερ θα μπορούσε να το απαντήσει, αλλά όντω δεν χρειάζεται το άρθρο αυτό για κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω, γιατί αυτό είναι μια συνήθις αναφορά παροχή μάλλον των στατιστικών στοιχείων προς την Eurostat. Θα έπρεπε να δηλαδή να είναι αναπόσπαστο τμήμα της ε, συνήθους ροής πληροφοριών προς την Eurostat. Ευχαριστώ, απλώς ήθελα να το ελέγξω. Κύριε Ρόντεμάχερ, θέλετε τώρα εσείς να απαντήσετε. Για το μορατόριο που ρωτήσατε ή για τα καθαρά σε δεδομένα. Ε, από όσο αντιλαμβάνομαι εγώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα έχουμε ε, προχωρήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με το σκεπτικισμό που δείχνετε εσείς. Υπάρχει πληθώρα κανόνων στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Ε, κανόνες ε, για ε, επανατιτλοποίηση, για ε, εταιρικές σχέσεις δημόσιο-οικονομικό τομέα, για τα SPVs, για τα swaps. δηλαδή, από όσο γνωρίζουμε, καλύπτουμε όλα τα πιθανά παραθυράκια, όλες τις πιθανές τρύπες, με το που προκύπτει η ανάγκη. Βέβαια χρειάζεται και ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη για ε, όλες αυτές τις συναλλαγές. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να ταξινομήσουν ή να επαναταξινομήσουν τα στοιχεία. Ε, Παραδείγματο χάρη για το 2001, άμα δεν υπήρχαν κανόνε, έτσι. Ε, με το που αλλάζουν οι κανόνε το 2008 και ισχύει ακόμη το χρέο, πρέπει να αναταξινομηθεί και να μπει στο δημόσιο τομέα. Το μορατόριο που ζητάτε λοιπόν είναι στο χρόνο και ήδη το, ε, το έχουμε συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιό μας. Ε, γιατί το σύστημα βάσει των ταμιακών ροών. Δεν ξέρω για ποια χώρα μιλούσατε. Υπάρχει μία χώρα που λειτουργεί με τέτοιους λογαριασμούς, ε, κυρίως όταν μιλάμε για τον κρατικό ισολογισμό, αλλά γίνεται προσαρμογή και μεταφέρουμε τις ε, καταχωρήσεις ε, ε, με βάση το σύστημα ταμιακών ροών και τις μετατρέπουμε σε καταχωρήσεις δεδουλευμένων. Η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών δεδομένων στο τομέα του χρέους και του ελλείμματος είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας πολύ υψηλότερη σε σχέση με τα άλλα 300 περίπου είδη στατιστικών στοιχείων που εκπονεί η Eurostat. Έχουμε ήδη σημειώσει δηλαδή μεγάλη πρόοδο. Uh, Σας ευχαριστούμε. Ε, κανείς ε, δεν ζητά να κάνει επερώτηση. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε, πιστεύω, το πρώτο τμήμα της ε, ακρόασής μας με κάποια ε, καθυστέρηση. Ελπίζω να μην δημιουργήσει προβλήματα η καθυστέρηση για το δεύτερο τμήμα. Ε, θα περάσουμε τώρα στο πάνελ εκπροσώπων ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παρακαλώ, ε, ελάτε στις θέσεις του Επιτρόπου και του κυρίου Ράντεμάχερ. Όσο αλλάζουν θέσεις θα ήθελα να πω κάτι, ίσως σας ξαφνιάσω ή ξαφνιάσω κάποια μέλη του ακροατηρίου ή και μέλη της Επιτροπής λέγοντας πως ε, κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα προσόντα επενδυτικών τραπεζών για να διαχειριστούν το χρέος τους. Ε, κανονικά δεν θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει αυτό Και στα πλαίσια του δεύτερου πάνελ μπορούμε να δούμε τις ε, κινητήριες δυνάμεις ε, ε, αυτής της επιχείρησης εκτός ισολογισμού. Τι κοστίζει να ακολουθήσει κάποιος αυτή την άγουσα και τι αν ακολουθήσει κάποια άλλη ρότα ε, τι είδους πιέσεις ασκήθηκαν ναι, για να δρομολογηθεί επιτυχώς το ευρώ και ε, ποιες πιέσεις υπήρξαν ε, για να είναι αξιόπιστο το σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή χρειάστηκε για να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας για τις κεφαλουχικές απαιτήσει να χρησιμοποιήσουμε συναλλαγές εκτός ισολογισμού ή υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος. Επίσης δημοσιεύματα σχετικά με ε, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και τις συμφωνίες ανταλλαγής αθέτηση υποχρεώσεων, δηλαδή τα credit default swaps. Επίσης ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία, το θεματοφυλάκιο ETCC, μπορούμε να διευκρινίσουμε αν υπήρξαν ε, υπερβολές σε σχέση με τις οικονομικές ε, μονάδες ε, όπως παραδείγματος χάρη τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα περίφημα hedge funds και αν έχουν δραστηριοποιηθεί άλλα λιγότερο ή περισσότερο νόμιμα κεφάλαια θα ακούσουμε παρουσιάσεις τώρα. Θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις στον Τζέραλτ Κόριγκαν που είναι ο διοικητής της Goldman Sachs Bank ε, των ΗΠΑ και πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ και μπορεί ίσως να μας δώσει κάποιες απαντήσεις και κατόπιν θα ακούσουμε τον Ρίτσαρτ Μέτκαλφ που είναι επικεφαλής της Παγκοσμίου Πολιτικής της ε, Διεθνούς Ενώσεως για τις Συμφωνίες Ανταλλαγής και τα παράγωγα ε, μπορεί να μας δώσουν μια σφαιρική εικόνα του κλάδου. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κόριγκαν. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και καθιστός μπορείτε να τα πείτε αν θέλετε, λέει η Πρόεδρος. Να είσαστε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση. Σήμερα το απόγευμα, όπως ξέρετε, υπάρχει και μια γραπτή δήλωσή μου προς την Επιτροπή σας, η οποία εστιάζεται στα θέματα αυτά της ε, ορθής διαχείρισης και της εποπτείας των χρηματαγορών. Για να είμαι σύντομος, θα σταθώ μονάχα στα κύρια σημεία αυτής της δήλωσης και δεν θα μπορώ να διαβάσω όλο το κείμενο. Το πρώτο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονίσω ήταν σαφές νομίζω από την προηγούμενη συζήτηση. Είναι το θέμα λοιπόν της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και θα πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε ότι και στην περίπτωση των ιδιωτικών εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει σωστή ε, παροχή αναφορών. Βέβαια αυτό δεν είναι επιστήμη, είναι περισσότερο κοντά σε μια τέχνη. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στον οικονομικό τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποιες χρηματοοικονομικές ενέργειες οι οποίες δεν απεικονίζονται πλήρως στον προϋπολογισμό των χωρών αυτών. Για μένα αυτό είναι από τους, ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό να υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς όπως η Eurostat, το Congressional Budget Office, το γραφείο του προϋπολογισμού δηλαδή στις Ηνωμένες που είναι ανεξάρτητη φορείς για την λειτουργία των λογιστικών προτύπων και την εφαρμογή τους. Τώρα, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια σειρά από προκλήσεις σε ό,τι αφορά την διαχείριση του χρέους και ιδίως σε ό,τι αφορά το κρατικό χρέος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν μερικές κεντρικές αρχές οι οποίες να διέπουν στην διαχείριση του κρατικού χρέους. Θα αναφέρω μονάχα μερικέ από αυτέ, ε, τι άλλε θα τι βρείτε στη γραπτή μου παρουσίαση. Καταρχήν, θα πρέπει η διαδικασία διαχείριση του χρέου να αναγνωρίζει ορισμένα βασικά στοιχεία τη πραγματικότητα. Έχουμε δει περιπτώσει όπου οι χρηματαγορέ, ακόμα και η κοινή γνώμη, είναι έτοιμοι για κάποιο χρονικό διάστημα να δώσουν το ωφέλιμα τη αμφιβολίας σε ορισμένε χώρε, οι οποίε έχουν μεγάλα ελλείμματα στον προπολογισμό του. Αν παραμείνουν όμως και διαιωνίζονται αυτά τα ελλείμματα ή ακόμα περισσότερα αν διωγγώνονται, κάποια στιγμή χάνεται η ανοχή των αγορών και εξαφανίζεται. Όταν συμβαίνει αυτό, το κόστος αντιμετώπισης της, αξιο... της εξυπηρέτησης του χρέους ανεβαίνει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι φορείς όπως η Eurostat πρέπει να απολαμβάνουν ενός υψηλού βαθμού πολιτικής ανεξαρτησίας θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η πολιτική ανεξαρτησία με τις απαραίτητες ικανότητες της Eurostat είναι εξίσου σημαντική όπως και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μια περαιτέρω αρχή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρέους προφανώς είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιήσει κανείς το μείγμα των διαρκειών των χρεών των ομολόγων τα οποία εκδίδονται ακόμα και όταν αυτό είναι πολύ δάπανο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον τομέα αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει προσφυγή στις συμβουλές των εμπειρογνώμων της ιδιωτικής αγοράς και των χρηματαγορών για το ποια είναι η καλύτερη στρατηγική και τακτική για τη διαχείριση του χρέους. <clears throat> Γι' αυτό οι περισσότερες χώρες έχουν μια ομάδα των λεγόμενων primary dealers, δηλαδή των κυρίων συναλλασσομένων ε, τραπεζικών και πιστοντικών φορέων σε ό,τι αφορά τα κρατικά ομόλογα. Κάτι ακόμα το οποίο αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση είναι το γεγονός ότι τα πρότυπα λογιστικής και παροχής εκθέσεων σε ό,τι αφορά το κρατικό χρέος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διάφανα αυτά τα πρότυπα και θα πρέπει εν καιρό να προσπαθούν να επιτύχουν μια συνεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή να είναι συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία. Βλέπω να υπάρχει μια κίνηση για μεγαλύτερη εναρμόνιση σε διαμεθοριακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις γενικές κατευθυντήριες αρχές και τις ε, αρχές σε ό,τι αφορά τις ε, αναφορές και τις εκθέσεις για το δημόσιο χρέος και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν πρόκειται να λύσουν αυτές οι αρχές όλα τα προβλήματα. Όταν υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν ελλείμματα, πρέπει κανείς να τα χρηματοδοτεί αλλά στο βαθμό που τηρεί κανείς αυτές τις αρχές μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ανοιχτή και ανθεκτική αγορά που θα παρέχει χρηματοδότηση στις, στους κρατικές οντότητες. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι σημαντικό να σταθούμε και στο θέμα της εποπτείας των ε, χρηματοοικονομικών παραγόγων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ πλοκό θέμα, αλλά θέλω να τονίσω Καταρχήν, ότι παρά τις δύσκολες περιστάσεις που περάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος ξεκινώντας από το 2005 για να αντιμετωπίσουμε τις λεγόμενες κόκκινες σημαίες. Θέματα λοιπόν που είναι στοιχεία αδυναμίας των υποδομών στις χρηματαγοράς. Αυτές οι κόκκινες σημαίες πολλές φορές έχουν ε, αναρτηθεί από ομάδες του χρηματοοικονομικού κόσμου. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η Τράπεζα της Federal Reserve της Νέας Υόρκης και η Διεθνής Κοινότητα των Κεντρικών Τραπεζών και αυτό περιλαμβάνει και αξιωματούχους από την Ευρώπη και χάρη σε όλες αυτές τις ενέργειες και τη συνεργασία έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος τα τελευταία πέντε χρόνια για να μπορέσουμε να μειώσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαδοτικές αδυναμίες των συστημάτων και θα έλεγα ότι χωρίς αυτές τις πρωτοβουλίες η χρηματοοικονομική κρίση στην οποία διερχόμαστε θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερη, ακόμα πιο δύσκολη για να αντιμετωπιστεί. Αναφέρω στην γραπτή μου δήλωση πέντε ή έξι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες βοηθούν την αντιμετώπιση της ε, κρίσης. Δεν πρόκειται να τα αναφέρω όλα αυτά, μόνο την τελευταία θα αναφέρω ότι μετά από παρατεταμένες συζητήσεις μεταξύ των ε, συμμετεχόνων στην αγορά των ρυθμιστών και διάφορους φορείς επαγγελματικούς, υπάρχουν πια οι κεντρικοί φορείς, κεντρικές διευκολύνσεις μάλλον συμψηφισμού μεταξύ αντισυμβαλωμένων σε ό,τι αφορά τα διάφορες μορφές συναλλαγών, παραδείγματος χάρη για τα credit default swaps, για τα CDS, δηλαδή συμφωνίες ανταλλαγής αθετήσεως υποχρεώσεων με την καινοτομία αυτή έχει μειωθεί σημαντικά ο συστημικός κίνδυνος ο οποίος συνάπτεται με την εμπορία παραγόγων ιδίως σε ό,τι αφορά τα CDF, τα swaps. Αλλά πρέπει να τονίσω επίσης και το συνοψίζω εδώ σε σχέση με το κείμενό μου υπάρχουν δύο ακόμα ή τρεις ακόμα σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Καταρχήν, το να υπάρχει κεντρικός συμψηφισμός σε όλα τα προτυποποιημένα παράγωγα μεταξύ ε, εμπόρων στις χρηματαγορές και των άλλων συμμετοχών στην αγορά, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο έγκαιρη πληροφόρηση όλων. Αυτό είναι πολύ θετικό και θα πρέπει να τονίσω στα πλαίσια αυτά, στο πλαίσιο αυτό ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, περίπου 95% των θέσεων για τα swaps που είναι ανοιχτές, και πολλές μη πρότυπες και μη καλυπτόμενες ηλεκτρονικά θέσεις καταγράφονται στην ε, εταιρεία αυτή, στον φορέα αυτό, ο οποίος καταγράφει τις προς θέσεις σε, ε, σε παράγωγα και μια παρόμοια ρύθμιση προβλέπεται για τα παράγωγα επιτοκίων και τα παράγωγα μετοχικού χαρακτήρα. Επομένως, θα είναι δυνατόν μέσω των ε, εβδομαδιαίων εκθέσεων αυτού του φορέα για την καταγραφή των συμψηφισμών να υπάρχει πράγματι πληροφορία για τα swaps και αυτό φυσικά θα περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία αφορούν κυρίαρχα κράτη και το χρέος κυριάρχων κρατών. Τέτοια μέτρα λοιπόν και επίσης όλη η συμμετοχή των ε, εμπλεκομένων στις διαδικασίες εκτός αγοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε πιο αυστηρές προϋποθέσεις σε σχέση με κεφάλαιο και σε καλύτερη προληπτική εποπτεία από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα η προληπτική εποπτεία σε όλες τις χώρες έχει την ικανότητα να απαιτήσει πληροφορίες σε σχέση με συναλλαγές, στοιχεία σε σχέση με την έκθεση των θέσεων των εταιριών αυτών και άλλες πληροφορίες βάσει της κρίσης των ρυθμιστικών αρχών. Και από την άποψη αυτή, οι έρευνες από τις ρυθμιστικές αρχές που αφορούν σε προβλήματα με την εγκυοδοσία ή με ε, περιθώρια τα οποία εφαρμόζονται σε γυμνή πώληση ε, αξιογράφων μπορούν να βοηθήσουν να εντοπίσουμε προβλήματα τα οποία αναδύονται. Τέτοιου είδου λοιπόν πρωτοβουλίε μαζί με άλλα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί, κατά την άποψή μου, είναι και αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την διαφάνεια της αγοράς παραγόγων εκτός αγοράς, over the counter δηλαδή. Αλλά μέσα στα πλαίσια αυτών των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να εξασφαλίσουμε ότι οι αγορές αυτές over the counter εξακολουθούν να παίζουν το σημαντικό τους ρόλο για την παροχή ε, ρευστότητος και καθορισμού τιμών τόσο στον τομέα των ε, παραγωγών όσο και στον, σε ό,τι αφορά την αγορά ρευστού για ένα μεγάλο πλαίσιο χρηματοδοτικών εργαλείων που παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην σύνολη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όποιος... Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον ε, δεύτερη παρουσίαση από τον Ρίτσαρντ Μέτκαλφ. Οι διάφοροι συνάδελφοι ήδη έχουν αρχίσει να ζητούν το λόγο. Κρατήστε την όρεξή σας να ακούσουμε και τον κύριο Μέτκαλφ. Σας ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Εγώ θα εστιάσω στο θέμα της οικονομικής και δημοσιονομικής διαφάνειας. Τα θέματα κλειδιά είναι η στεναρότητα των υποδομών και η βελτίωση στην ε, διαχείριση κινδύνου των αντισυμβαλωμένων. Πιστεύω πως ε, είναι ένας τομέας όπου εμείς ως κλάδος μπορούμε να συνεργαστούμε παραγωγικά με την νομοθετική εποπτική κοινότητα ε, γιατί ρητό μας είναι ότι το φως του ήλιου είναι το καλύτερο αντισηπτικό. Θα σας πω βέβαια ότι επειδή δεν έχουμε ε, εντολή, δεν είναι μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες να πούμε τι είδους αναφορά είναι για η ε, κατάλληλη ή προς ποιον. Ε, περισσότερο εγώ θα μιλήσω για την ακυρεότητα της αγοράς όσον αφορά τα παράγωγα OTC. Η διαφάνεια για την υπόλοιπη αγορά και αυτό είναι ξεχωριστό θέμα το οποίο απαιτεί μια ανάλυση κόστους ωφέλειας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω από αυτού του θέματος είναι ότι κατά ε, σε μόνιμο βάση βλέπουμε πως η διαφάνεια φαίνεται να ακολουθεί την εξέλιξη της ρευστότητα. Δεν είναι αντίστροφα τα πράγματα. Ως εμπορικός σύνδεσμος αντιπροσωπεύουμε ένα πλήρη, ε, πλήρες φάσμα διαφόρων ε, οργανισμών, ακόμα και κυριάρχων κρατών. Έχουμε περίπου 820 ε, ε, μέλη ε, και χρησιμοποιούν τα OTC για να διαχειριστούν τους κινδύνους και το κάνουν αυτό από τις αρχές του 1980. Δηλαδή αυτά τα μέσα δεν είναι και τόσο φνέα. Η πρώτη περίπτωση παραγόγων ήταν μια ανταλλαγή σε ρευστό με την Παγκόσμια Τράπεζα. θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη ανάπτυξη όσον αφορά τα λογιστικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την αγορά. Αυτό που πιστεύουν όλα τα μέλη μας σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα, όπως σας είπα, μελών, τονίζουν πως η εποπτική διαφάνεια μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, πράγμα το οποίο θα εξυπηρετήσει και την οικονομία. Εκεί όπου το θέμα, η αγορά είναι σημαντική και συστημικά σημαντική, θα πρέπει να είναι σαφές πως ο όγκος κινδύνου μέσω των συμβάσεων παραγόγων είναι μόνο ένα κλάσμα των όσων συμβαίνουν στις ε, αγορές τίτλων, δηλαδή μετοχές, ομόλογα κτλ. Δεν είναι και τόσο κοινό το φαινόμενο και παρομοίω τα ποσά αυτά είναι μόνο ένα ε, απειροελάχιστο κλάσμα του ΑΕΠ. Νομίζω πω η διαφάνεια τη εποπτείας μπορεί να επιφέρει δύο βασικά ωφέλη. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να αποφύγουμε τι ε, δυνατότητε χειραγώγηση τη αγορά, Όσο σπάνιο και αν είναι αυτό, υποβαθμίζει και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην αγορά και την εμπιστοσύνη των ε, συμμετεχόντων στην αγορά και το δεύτερο στοιχείο είναι η συστημική εποπτεία, δηλαδή η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πιθανή σώρευση ε, λανθασμένων θέσεων είτε σε ολόκληρη την αγορά είτε μέσω μάλλον από πλευρά μια και μόνη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει δυνητικά υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο. Αυτή η στόχη είναι κοινή και για τον κλάδο μας γιατί φυσικά βλάπτουν τις επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει εποπτεία βέβαια δεν υπάρχει λόγος η αγορά να μην μπορεί να λειτουργεί ελεύθερα μέσω ενός μεγάλου εύρους συμβάσεων που χρησιμοποιούνται από την σύγχρονη οικονομία. Επίσης είναι σαφές ότι οι λύσεις στα θέματα ακαιρεότητας αγοράς είναι σχετικά απλές, τουλάχιστον όσον αφορά την σύλληψή του. Δηλαδή, αναφορά των συναλλαγών, αναφορά των παθητικών πολύ, πολύ κοντά στην πραγματικό χρόνο. Ένα παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που ήδη έχει ένα ευρύ καθεστώς καταγραφής των συναλλαγών πέρα από τις απαιτήσει της ΜΕΦΕΤ. Το να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα σημαίνει επόπτες που πρέπει να διακρίνουν από τη μια πλευρά την αληθινή και σωστή διαδικασία σχηματισμού τιμών, όπου παίζουν σημαντικό ρόλο τα παράγωγα γιατί διασφαλίζουν μια αμφίδρομη αγορά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε έτσι διαπιστώνονται οι καταχρηστικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να στρεβλώσουν τις τιμές και στις δύο περιπτώσεις είναι ζωτική σημασία σε υποπτία και όσον αφορά την συστηματική ε, γενική εικόνα τα μητρώα στοιχείων ε, για τις εμπορικές συναλλαγές δίνουν ε, στοιχεία για όλες τις τάξεις παραγόγων αλλά και στοιχείων ενεργητικού. Όλα τα στοιχεία δηλαδή συλλέγονται σε συγκεκριμένο σημείο, όπως γίνεται ας πούμε για τις πιστώσεις ή για τις μετοχές. Επειδή η έκθεση των συμβαλωμένων μερών μπορεί να σωρευτεί και διασυνοριακά, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείται μια ε, ε, ομαδοποιημένη ε, εικόνα, σφαιρική εικόνα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μόνο ένα ενιαίο μητρό, όχι μόνο γιατί είναι πιο φθηνό για την αγορά, αλλά γιατί βελτιώνει τα στάνταρ αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Φυσικά κάποιες από τις λεπτομέρειες που εντάσσονται στην διασφάλιση της αναφοράς των συναλλαγών μπορεί να είναι κάπως δύσκολα στην εφαρμογή. Θα πρέπει να έχουμε τεχνικές προδιαγραφές και μια συγκεκριμένη γλώσσα αναφοράς. Ευτυχώ κάποια από αυτά ήδη υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κάποιες νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του πελάτη, όσον αφορά τις συναλλαγές σε παράγωγα. Και εκεί και η αγορά είναι πρόθυμη να δώσει τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν νομικά εμπόδια σε κάποιε δικαιοδοσίε. Και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε στενά με του επόπτε, ώστε να καθορίσουμε την κλίμακα αυτή τη πρόκληση, αλλά και το... τι πιθανέ λύσει που μπορούμε να βρούμε. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η πηγή στην περίπτωση ε, παραγόγων πιστώσεων Μα δίνουν σημαντικές πληροφορίε όσον αφορά την ομαδοποιημένη κλίμακα παραγόγων. Τα στοιχεία της, της DTCC δημοσιεύονται εβδομαδιαία και δείχνουν ότι αυτές οι θέσεις είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού τζίρου και πολύ μικρό ε, ποσοστό των εκκρεμών ε, δανείων. Των εκκρεμών των δανείων. οι δημοσιονομικές ροές φαίνεται να γίνονται στο μεγαλύτερο, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μέσω χρεογράφων. Στον τομέα των πιστώσεων όπως ε, των δανείων, όπως έχουμε πει και προηγουπτήτερα για τα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης, αυτά ανέρχονται μόνο στο 2% των εκκρεμών, ε, εκκρεμών των δανείων. Ταυτόχρονα για τους μεγάλους επενδυτές που χρησιμοποιούν ε, τα CDS η διαθεσιμότητα αυτών των μέσων τους δίνει τη δυνατότητα περισσότερη εμπιστοσύνη για να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και σίγουρα ο περιορισμός της χρήσης των CDS θα οδηγούσε αυτούς τους επενδυτές να ζητούν μεγαλύτερη απόδοση ώστε να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα. Και αυτό φυσικά αυξάνει το κόστος του δανεισμού με τη σειρά τους. Σε διεθνή, είμαστε διεθνής ε, ένωση με μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο και 23 από τα 27 κράτη και υποστηρίζουμε την εποπτεία των εισαγορά των παραγόγων και κατά συνέπεια θεωρούμε πως μια ρεαλιστική προσέγγιση στα θέματα τοποθεσίας και υποδομών θα είναι πολύ σημαντική. Και αυτό λόγω της φύσης των αγορών ο διασυνοριακός συντονισμός είναι πολύ σημαντικός και αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε συστημική εποπτεία κινδύνου δεν υπάρχει άλλη υπεύθυνη εναλλακτική λύση από τον διεθνή συντονισμό. Και επίσης, με παρόδο για το θέμα των μεγά, της μεγάλης έκθεσης, ε, υποστηρίζουμε το, και παρακολουθούμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτήσει νομοθεσία με, μέσα, μέτρα μάλλον τα οποία απευθύνονται περισσότερο στην μεγάλη έκθεση. Πιστεύουμε πως ε, η πειθαρχία στους λογαριασμούς market to market είναι πολύ σημαντική γιατί αυτό οδηγεί και τα φέρνει τα παράγωγα στους ισολογισμούς. Ίσως λοιπόν χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά, κάποια πολύ δύσκολη, κάποια πιο τεχνική, κάποια που εξαρτάται μόνο από την πολιτική βούληση και συμφωνία. Ωστόσο θεωρούμε πως έχουμε κοινό προορισμό και όπως είπα και προηγούμενα, αν ε, χρειαζόταν να συνοψίσω, ε, όπως σας είπα, το φως του ήλιου είναι το καλύτερο αντισηπτικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών που είναι ακόμη εδώ. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους κάποιων μελών, αλλά πρέπει να επιστρέψουν. Schmidt and Werner Langen. Um, so we'll start with Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις δύο αυτές ε, παρουσιάσεις. Ε, μιλώντας εις βάθον για το θέμα των παραγωγών και για το, τη μελλοντική ρύθμιση του κλάδου, λαμβάνουμε ενθαρρυντικά μηνύματα. Όμως, το να ασχολούμαστε με τα παράγωγα εκτός αγοράς και το κεντρικό συμψηφισμό δεν νομίζω ότι επαρκεί για να επιλύσουμε τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος Κόριγκαν ε, στην πρώτη παρουσίαση. Ξέρω ότι δεν είναι στη μόνη τράπεζα που τιτλοποίησε χρέος ε, για ε, κυρίαρχα κράτη. Πολλοί από τους συναδέλφους σας τα ίδια κάνανε θα ήταν χρήσιμο και ας ξεπερδέψουμε αυτή την πρώτη ερώτηση. Χρησιμοποιώντας ε, τα swaps ε, δημοσίων ε, χρεών, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα χρηματοπιστωτικό παράγωγο που πωλείται υπέρ του κράτους και ένα παράγωγο που πωλείται για να κρύψουμε ένα χρέος. Και ποιος είναι υπόλογος, αυτός που το πουλάει ή αυτός που το αγοράζει. Ε, και το duty of care το περίφημο, ε, δηλαδή ποιος έχει την ε, ευθύνη, ποιος πρέπει να υπομειστεί την ευθύνη. Αυτό θα μας βοηθούσε να μάθουμε. Αυτό μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το απαντήσετε. Κυρία Ποδηματά, θα ακούσουμε την ερώτηση κυρίας Ποδηματά και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο εισηγητές για τις ε, παρεμβάσεις τους. Το ερώτημά μου αφορά σε μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου από τον, τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδος και του Λουξεμβούργου, την Γερμανίδα Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, εδώ είμαι, και τον ε, Πρόεδρο της Γαλλίας, οι οποίοι με κοινή του επιστολή στον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, ζήτησαν να διεξαχθεί κάποια έρευνα για το ρόλο και τις επιπτώσεις της κερδοσκοπίας στα συμβόλαια διασφάλισης κινδύνου στα CDS επικρατικών ομολόγων, συγκεκριμένα των ελληνικών κρατικών ομολόγων και παράλληλα ζήτησαν να ενισχυθεί η ασφάλεια των αγορών εξωχρηματιστηριακών παραγόγων ε, με την ε, θέσπιση με τη συγκρότηση ενός ε, κεντρικού αντισυμβαλόμενου για την, εκαθάριση για το διακανονισμό. θέλω να σας ρωτήσω πώς νομίζετε ότι μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία μιας τέτοιας οντότητας με τη δημιουργία της οποίας αντελήφθηκα από τις σημερινές σας παρεμβάσεις ότι συμφωνείτε; επίσης εάν συμφωνείτε ότι πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα όρια ε, διακράτησης στην εμπορία των cds όπως προτείνεται με την ε, συγκεκριμένη επιστολή και ότι τέλος εάν πρέπει να απαγορευτούν οι κερδοσκοπικές συναλλαγές cds να απαγορευτεί δηλαδή η απόκτηση cds που δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Κόριγκαν, θέλετε να απαντήσετε πρώτος και μετά ο κύριος Μετ Καλφ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση εδώ για την κυρία εκ δεξιών. Υπάρχουν και άλλες βέβαια. Ε, μιλήσατε για απόκρυψη. Ε, ας μην το παρακάνουμε, ας μην υπερβάλλουμε. Δεν νομίζω ότι ενδείκνυται ο όρος για να περιγράψουμε κάποιες καταστάσεις στις οποίες ε, αναφέρεστε. Τώρα αν υπάρχει υπερβολική ε, απόκρυψη αυτό είναι άλλο θέμα. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε χρειαζόταν μεγαλύτερη διαφάνεια. Επ' αυτού θα συμφωνήσω μαζί σας. Ε, και μην ξεχνάτε ότι οι εν λόγω συναλλαγές ανάμεσα στην Goldman Sachs και την Ελλάδα ε, ε, έγιναν πριν από μία δεκαετία. Χρειάζεται διαφάνεια για την κοινοποίηση των πληροφοριών, συμφωνώ. Αλλά νομίζω άλλο ρωτήσατε. Αν θεωρώ ότι οι δυνατότητες ε, διαφάνειας ε, μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή για την καταγραφή του χρέους και για το χαρακτηρισμό κάποιων συναλλαγών και για τα δύο. αν μπορούν να εφαρμοστούν για τον αγοραστή και για τον πολιτή και ποιος φέρει την ευθύνη. Και οι δύο είναι η απάντηση. θα έπρεπε ίσως γραπτός να γνωρίζουμε ποια είναι η απόλυτη και ποια η σχετική ευθύνη και του αγοραστή και του πολίτη. Από τη δική μου εμπειρία θα έλεγα ότι μία από τις ευθύνες που έχουν κρίσιμη σημασία για τον πολιτή είναι να υπάρχει διαφάνεια ακόμη και αν ε, οι πελάτες μεριμνούν ώστε η τεκμηρίωση των συναλλαγών ε, ε, είναι πλήρης και κατανοητή. Τώρα, υπέροχο αυτό το ερώτημά σας, ποιος είναι υπεύθυνος και τονίζω και οι δύο είναι υπεύθυνοι. Ε, όσο το έχουμε κατά νου, νομίζω, καλά πάμε. Δεύτερη ερώτηση. Αυτός ο όρος, ο άλλος όρος, κερδοσκοπία, ε, ε, είναι πολύ βεβαρημένος ο όρος αυτός χρησιμοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Αυτός ο όρος λοιπόν, κερδοσκοπία και πώς τον βλέπουμε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι απλή έννοια, αλλά και φευγαλέα ταυτόχρονα. Στην αγορά παραγωγών και στις άλλες, τι συμβαίνει. Για κάθε αγοραστή υπάρχει πολιτή και για κάθε πολιτή, ε, για πολιτή υπάρχει αγοραστής. Έτσι δουλεύουν οι αγορές. Αν θέλει κάποιος μία επιχείρηση ή ένα κράτος να κάνει μία συναλλαγή, χρειάζεται κάποιος στην άλλη άκρη. Απαραίτητα. Ε, ε, εξετάστε το με προσοχή αυτό που σας λέω. Ε, σε αυτή την δυναμική των long και των short, των ακάλυπτων και των καλυμμένων πωλήσεων υπάρχει και το θέμα του συμψηφισμού κάθε φορά για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Ε, καταλαβαίνω αυτά που είπατε για, τη, για τα όσα εμπεριέχει η δήλωσή μου. Αλλά τι θα έλεγα. Όταν μιλάμε παραδείγματο χάρη για ένα μηχανισμό κεντρικής εκαθάρισης, για να μιλάμε για την ουσία, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να είναι ρυθμισμένος ο μηχανισμός και πρέπει να υπάρχει ε, επαρκή αυστηρότητα. Δηλαδή πρότυπα σχετικά με το ποιο μπορεί να είναι μέλο αυτών των οργανώσεων συμψηφισμού και ε, βάσει ποιων όρων μπορεί ε, να καθαιρεθεί ένα μέλος, να αποπεμφθεί. Αυτά τα επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια εγώ και το ξέρουν οι συνάδελφοί μου. Ας περάσω στα CCPs τώρα. Θα πρέπει να αποδειχθεί ε, στις ε, ρυθμιστικές αρχές ε, και μέσω των δοκιμών που γίνονται ότι αυτές οι κεντρικές αρχές συμψηφισμού των αντισυμβαλωμένων πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και πιστέψτε με ότι μόνο έτσι κατοχυρώνεται η χρηματοπιστωτική ακαιρεότητα. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για την ε, κερδοσκοπία, αλλά πραγματικά είμαι πλήρως πεπισμένος πως οι μεταρρυθμίσεις που τώρα γίνονται και κάποιες ε, που έχουν ήδη γίνει μπορούν να σας καλύψουν στην ερώτηση που υποβάλλατε και εξάλλου οι επόμενε εξελίξει που θα ακολουθήσουν τους προσεχείς 12 ή 18 μήνες σχετικά με την διαθεσιμότητα των πληροφοριών ω προ τις συναλλαγέ θα αυξήσουν τη διαφάνεια για τα κράτη, για τις επιχειρήσεις και για τις ρυθμιστικές αρχές ούτως ώστε όλοι να είμαστε, πώς να το πω, πιο καθησυχασμένοι σε σχέση με τώρα. Ευχαριστώ κύριο Μέτκαλφ. Για το πρώτο ερώτημα δεν ξέρω αν απευθύνονταν και σε μένα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Συμφωνώ ότι η ευθύνη είναι μοιρασμένη. Η μεγαλύτερη ευθύνη σίγουρα αυξάνεται όταν μιλάμε για λιανικό εμπόριο χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αλλά στην αγορά παραγόγων over the counter εκτός αγοράς δεν πρόκειται για λιανικό εμπόριο τέτοιων προϊόντων. Συνήθως έχετε κάποιο διαχειριστή ε, ενός κεφαλαίου, ενός ταμείου που χρησιμοποιεί τα CDS, τα swaps για να ασφαλίσει το χρηματοφυλάκιό του και ο οποίος δεν θα θέλει κατά ανάγκη να δώσει όλες τις πληροφορίες σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά. Αυτή είναι λοιπόν μια δυνατή απάντηση σε ό,τι αφορά τώρα τις έρευνες, την έρευνα για ενδεχόμενη κερδοσκοπική δραστηριότητα, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει καταρχήν ένα πρόβλημα καθορισμού του τι σημαίνει κερδοσκοπία. Παραδείγματος χάρη τα CDS, τα swaps. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα swap εκτός εάν οι δύο συμβαλόμενοι έχουν αντίθετες απόψεις σε σχέση με την κίνηση των αξιών στο μέλλον. Αυτή είναι η φύση της συμφωνίας. Ο ένας αγοράζει από τον άλλο προστασία, ο άλλος παίρνει ένα κέρδος επειδή παρέχει αυτήν την ασφάλεια και λέει ότι υπάρχει μια τιμή ασφαλείας για τα, για τα ομόλογα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το οποίο λέμε freelance. Δεν υπάρχει δωρεάν ασφάλιση γιατί κανείς πρέπει να πληρώσει κάτι για αυτή την ασφάλιση. Επομένως, κοντολογής είναι πολύ καλό να γίνει μια έρευνα για τη δραστηριότητα στις χρηματαγορές. Θα καταλάβει κανείς άμα κάνει αυτή την έρευνα ότι είναι πραγματικά μια υγιής αγορά η οποία όμως αρέσκεται στους κινδύνους για το ρόλο τώρα των φορέων συμψηφισμού μεταξύ αντισυμβαλωμένων, αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή. Υπάρχει συγκέντρωση θέσεων κινδύνου όταν δημιουργούνται κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσει κανείς ότι αυτή η αγορά είναι πράγματι εύρωστη και μπορεί να αντέξει την πτώχευση, την, την αδυναμία εξυπηρέτησης από ένα μεγάλο μέρος της. Εμείς έχουμε δει ότι η διμερής, το διμερές netting, ο διμερής συμπληφισμός έχει πράγματι να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαδικασία της Lehman Brothers, ιδίω όταν αφορά και την αντιμετώπιση των εγγύσεων, κάτι το οποίο είναι πολύ ρουτίνας θέμα και πρόβλημα σε τέτοιου είδους δοσοληψίες μεταξύ οικονομικών φορέων. Θέλει κάποιος άλλος να συνεχίσει, λέει η πρόεδρος. Ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν και μετά ο Νικόλας Θανησίους. Χάνς Πέτερ πρώτα. Κύριε Κόριγκαν, πάντα είναι κάτι το οποίο μας δίνει ιδέες και μας εμπλουτίζει να είμαστε σε επαφή με εκπροσώπους Goldman Sachs είτε στην Νέα Υόρκη, είτε στην Αυστραλία, είτε στη χώρα μου, την Αυστρία. Εμείς αναρωτιόμαστε και είμαστε εντυπωσιασμένοι για την επιτυχία της εταιρείας σας τα τελευταία χρόνια, για, τα, για την πολύ καλή της απόδοση. Άλλες εταιρείες έχουν μπατήρι και εσείς τα έχετε καταφέρει πολύ καλά στον τομέα αυτό τον επενδυτικό. Αν υπήρχε μία δυνατότητα να δεχτείτε μία προσφορά από την ελληνική κυβέρνηση και να ασχοληθείτε με την διαδικασία των swap, των υπολογισμών των swap σε σχέση με την Ελλάδα, με την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Θα το ξανακάνατε, η Goldman Sachs θα ξαναέμπαινε σε ένα τέτοιο παιχνίδι ή θα λέγατε ότι αυτό ήταν αρνητικό για τη φήμη σας. Και ένα άλλο γενικό ερώτημα. Συμφωνείτε με τους παρατηρητές που λένε στο σημερινό κόμμα κόσμο ότι η Goldman Sachs έχει μεγαλύτερη εξουσία από τον Πάπα. Ε. We can't δεν ακούσαμε τι είπατε. Σε λίγο θα σας δώσω και τις ε, λεπτομέρειες. Αλλά να σας πω ότι ακόμη και ο Πάπας έχει προβλήματα τη σήμερον ημέρα. Αυτό προς το παρόν. Εκτός από τον Πάπα είχε προβλήματα και ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ξέρετε, ο οποίος εφλέρταρε μια νεαρή κυρία της εποχής και της είπε εκ γυναικός προκύπτει τα φαύλα. Του απήντησε η έξυπνη αυτή κοπέλα τότε ότι και εκ γυναικός προκύπτει τα κρίτο, τα καλύτερα. Χάλασε το ειδήλιο. Θέλω να πω το εξή ότι στη σημερινή εποχή από την Αμερική προκύπτουν τα φαύλα και από την Αμερική προκύπτουν τα κρίτο τα φαύλα είναι ότι μας δημιουργήσατε την κρίση και πρέπει να συμφωνήσετε, μας τη μεταφέρατε και στην Ευρώπη και τα κρίτο είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσετε να βγει και η Ευρώπη από αυτό το πρόβλημα που της δημιουργήσατε. Μετά από την παρένθεση αυτή θα θέλω να σας πω τα εξή. Αυτή τη στιγμή ένα στοιχείο που ξεπερνάει την κρίση οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής είναι ότι κόβει χαρτονόμισμα. Δεν κόβουμε χαρτονόμισμα εδώ στην Ευρώπη. Συνεπώ θα έπρεπε η ισοτιμία να πέφτει και θα έπρεπε η αξιοπιστία του νομίσματος εκείνου να είναι μικρότερη από την αξιοπιστία του ευρώ. Σας ερωτώ, δεν θα πρέπει εσείς σαν commercial bank, όχι σαν σε θεωρητικό επίπεδο να μας τα λέτε αυτά που τα μας τα είπατε τόσο ωραία θεωρητικά, να βοηθήσετε στην αποκατάσταση αυτής της οτιμίας και να πείτε στους πελάτες σας ότι είναι πιο ασφαλές το ευρώ το οποίο δεν κόβει καινούριο νόμισμα από ότι η Αμερική η οποία κόβει συνέχεια νόμισμα. Ευχαριστώ. Right. I'm not sure whether you're the Pope or a temptress, but um, δεν είμαι σίγουρος, ε, σίγουρη κύριε Κόρεγκαν ε, αν ε, είστε ο Πάπας ή απλώς ο πειρασμός, αλλά απαντήστε αν θέλετε. Ξαναγυρίζω εδώ. Αν αφήσουμε τον Πάπα στα προβλήματά του, το ερώτημα είναι γνωρίζοντας αυτά τα οποία ξέρουμε, αν αντιμετωπίζαμε τις ίδιες καταστάσεις όπως αυτές οι οποίες οδήγησαν στα, στις ε, συμφωνίες ανταλλαγής ε, συναλλαγμάτων το 1998 μέχρι το 2000 θα κάναμε τα ίδια πράγματα και πάλι. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσα να δώσω σε αυτό το ερώτημα θα ήταν να σας πω ότι δεν μπορεί κανείς να γυρίσει 10 χρόνια πίσω τη σημερινή αντιμετώπιση και σκέψη. Δεν υπάρχει καμιά σχεδόν αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ακόμα κι αν είχαμε ακριβώς τις ίδιες ταυτόσιμες συνθήκες σήμερα που φυσικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο θα το ξανακάνουμε κατά πάσα πιθανότητα αλλά θα το κάναμε κάπως διαφορετικό. Και με επαναφέρει αυτό στο προηγούμενο ερώτημα το οποίο προχωρά λίγο περισσότερο σε σχέση με το γεγονός ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η ευθύνη και του αγοραστή και του πολιτή. Θέλω να τονίσω καταρχήν ότι ακόμα και το 1998, 1999, 2000 ο κύριος στόχος, ο αρχικός κύριος στόχος των swaps αυτών που έγιναν με την Ελλάδα ήταν να επιτρέψουν στην Ελλάδα να μετατρέψει χρέος σε δολάριο, σε χρέος σε ευρώ. Γιατί αυτό ήταν το τίμημα του να γίνει μέλος της, ευρωπαϊκής, της ζώνης του ευρώ και να εισαγάγει το ευρώ ως το επίσημο νόμισμα στην Ελλάδα. Η λογική, επομένως, και η βάση αυτής της ε, απόφασης που ελήφθη από την Ελλάδα και την Goldman Sachs τότε ήταν αυτή. Ήταν μια απόλυτα φυσιολογική και ορθολογική βάση. Ήτανε, νομίζω ότι αυτό είναι αδιαφυσβήτητο ακόμα και αν γυρίσω πίσω 10 χρόνια, ο στόχος του να μπορέσει η Ελλάδα να μπει στη ζώνη του ευρώ. Τώρα, όταν έγιναν αυτά τα πρώτα swap, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα το οποίο τίθεται, περάσαμε μια χρονική περίοδο μέσα στην οποία το ευρώ ανατιμήθηκε σε σχέση με το δολάριο και το γεν σημαντικά. Και επομένως η άνοδος της τιμής του, του ευρώ εναντί του δολαρίου ήταν αναστροφή αυτή της ε, τάσης που είχε γίνει το 2000-2001 όταν έπεθε το ευρώ σε σχέση με το δολάριο που οδήγησε την Ελλάδα να κάνει αυτές τις ε, ανταλλαγές συναλλαγμάτων βασιζόμενοι σε ιστορικές αξίες της ισοτιμίας αυτής. Ήταν αυτή η ανάγκη και η ανάγκη να αναθεωρήσει, να αναδιαρθωθούν οι αρχικές ε, ανταλλαγές συναλλαγμάτων που οδήγησαν σε ανταλλαγή επιτοκίων μεταξύ Λάδος και Goldman Sachs, αυτά οδήγησαν στα προβλήματα τα οποία αναφέρεται εδώ. Γιατί <clears throat> αυτό το οποίο έγινε ήταν να διορθωθούν οι ισοτιμίες της ε, αγοράς που περιλαμβανόντουσαν στα, στα swaps και αυτό οδήγησε ουσιαστικά σε μείωση κατά 1,5% του δημοσίου χρέους της Ελλάδος σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Αλλά ακόμα και με αυτή την μικρή μείωση, το, η σχέση του χρέους προς το ΑΕΠ ήταν πάνω από 100%. Επομένως, για να απαντήσω και πάλι στο ερώτημα θα το επαναλαμβάνετε ή όχι, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι αν ισχύαν οι κανόνες οι οποίες ισχύουν τώρα μετά από το 2008 αν υπήρχαν αυτοί οι κανόνες που αναφέρονται για τη Eurostat, αν ισχύανε το 2001, θα είχε προκύψει τότε μια κατάσταση όπου τα χρήματα τα οποία χρωστούσε η Ελλάδα στην Goldman Sachs θα είχαν καταγραφεί μέσα στα πλαίσια του χρέους. Εμείς χρησιμοποίησαμε αν χρησιμοποιούσαμε λοιπόν τους κανόνες του 2008 στην περίπτωση αυτή, τότε δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να καταφύγει η Ελλάδα σε μια τέτοια ρύθμιση. Επομένως νομίζω ότι οι κανόνες του 2008 αλλάζουν την κατάσταση. Και δεν θα είχαμε και κανένα πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση να προβούμε σε μια νέα συναλλαγή αυτού του είδους. Τώρα, σε σχέση με το θέμα του ευρώ και του δολαρίου. Αυτό το οποίο λέτε έχει ένα μεγάλο μέρος αλήθειας. Ένα μεγάλο μέρος αλήθειας. Είναι πράγματι σημαντικά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου αλλά δεν ε, θέλω να διαφεσβητήσω ότι από πολλές απόψεις η πηγή της κρίσης προέρχεται από τις Ηνωμένε Και αν θέλετε να επεκτείνω το ερώτημά σας, σε σχέση με την ισοτιμία του δολαρίου και του ευρώ, μπορώ να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη καριέρα μου πριν από 25 χρόνια ως κεντρικός τραπεζίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα από τα πράγματα που έμαθα είναι ότι μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να καθορίζει τις πολιτικές ισοτιμιών. Επομένως, θα δεν θα σχολιάσω περισσότερο το ερώτημά σας. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και ο κύριος Μέτκαλφ. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να παρέμβουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, διευκρινήσεις. Μία επερώτηση θα κάνω. Είπατε ότι τότε οι συμφωνίες ανταλλαγής έγιναν σε τιμές αγοράς. Εγώ έχω τις εξής πληροφορίες. Η αξία του 2001 ήταν 2,4 δις ευρώ. Αυτή είναι μία, ένας ανελεκτικός τρόπος καταχώρησης του SWAP. Και στη συνέχεια το 2005... Υπάρχουν πληροφορίες ότι πουλήσατε το SWAP στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας για 5,1 δις. Έτσι αμφισβητώ αυτό που είπατε ότι το 2001 ήταν μια καθαρή τιμή αγοράς και σας ερωτώ υπήρχε κάποια κρυφή συνιστόσα μήπως βάσει της οποίας μειώθηκε το χρέος και ε, ανεστάλη ε, ε, ετεροχρονιστική για να καλυφθεί η είσοδος της χώρας στη ζώνη ευρώ. Απάντηση. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε μιλώντας για το 2005 και την πώληση στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας. Ε, αυτό που ξέρω είναι ότι οι περισσότερες εκθέσεις ε, που είχε η Goldman Sachs σε σχέση με την Ελλάδα για τον κίνδυνο πιστώσεων πωλήθηκαν σε άλλους παίκτες της αγοράς ε, το 2005. Δεν μπορώ να σχολιάσω στοιχεία που δεν γνωρίζω. Πάω πίσω τώρα στο 98, 99 και 2000-2001. Εγώ ε, κατανοώ εξής ε, τα δεδομένα. Το 98, δεν θυμάμαι και καλά, μπορεί να ήταν και το 99, η Goldman Sachs στην Ελλάδα άρχισε διάφορες συναλλαγές swaps συναλλάγματα και αυτές οι αρχικές συναλλαγές έγιναν σε τιμές αγοράς για ε, ξένα συναλλάγματα, για ξένα νομίσματα. Και έγινε σημαντική υποτίμηση κατόπιν το 2000 του ευρώ έναντι του δολαρίου και του γεν. Και υπό αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι, επανέλαβε δύο-τρεις ενδιάμεσες συμφωνίες ανταλλαγής και νομίζω ότι ήταν ε, στα τέλη του 2000, αν θυμάμαι καλά, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ε, τα ε, ιστορικά ε, ποσοστά ισοτιμίας που διαφέρουν λίαν από τα ποσοστά της αγοράς. Και σας θυμίζω ότι γινόταν με την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και του γεν. Οπότε, χρησιμοποιώντα αυτά τα στοιχεία, αυτή την εμπειρία, θα έλεγα ότι η χρήση όλων των εκκρεμών συμφωνιών ανταλλαγής ε, ε, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2001 οδήγησε σε αναδιάρθρωση των swaps χρησιμοποιώντας ιστορικούς συντελεστές ε, για την ισοτιμία. Και με την αναδιάρθρωση αυτή που έγινε χρησιμοποιώντας ε, τους ιστορικούς, ε, τις ιστορικές ε, ισοτιμίες οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή η αναδιάρθρωση τελικά είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η έκθεση της Goldman Sachs της Ελλάδος έναντι της Goldman Sachs βάσει των κανόνων που τότε ήταν αποδεκτοί και η υποχρέωση πώληση προς την Goldman Sachs εκειμενόταν στα 2,3-2,4 δις τότε. Οπότε, μείωση 1,5 ε, ε, ε, σε σχέση με το λόγο ΑΕ προς χρέος. και το χρέος 2,4 ε, προς την Goldman Sachs θα φαινόταν ως δάνειο αν χρησιμοποιούσαμε τους κανόνες ε, ε, ε ως χρέος συγγνώμη αν χρησιμοποιούσαμε τους κανόνες το 2008 ε, και δεν θα φαινόταν ως μείωση του λόγου του ΑΕΠ προς το χρέος. Ε, δεν μπορώ, ξέρετε, να ε, σχολιάσω τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποίησατε, αλλά εγώ αυτά θυμάμαι από εκείνη την περίοδο. So, Well. Θέλετε να... Ο κύριος, ναι, κύριος Ναι, συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Νόμιζα ότι αυτό που θέλατε να πείτε ήταν καλό να το ακούσουν και οι υπόλοιποι. Και ίσως θα έπρεπε να μείνει ο κύριο Ζαντεμάχερ για να ακούσει τη συνέχεια. Κύριε Μέτκαλφ, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Όχι. Όλοι Σμιτ, Πετ Λάγκερ, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας άκουσα, ε, κύριε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τους δύο. Ε, εγώ τα βρίσκω λογικά αυτά που λέτε. Ε, θα διαφωνήσουν κάποιοι συνάδελφοι, πάντως... Ε, δημόσιος ε, είστε στο εδόλιο. Δεν είναι αποδεκτές οι πρακτικές σας. Θα ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται να χάσετε ε, την αξιοπιστία σας. τι μπορείτε να κάνετε για να, να στρέψετε την απώλεια της πίσης κοινής γνώμης σε εσάς ούτε λίγο δεν σας πιστεύουν σήμερα, ξέρετε. Καλό είναι αυτό που, αυτά καλά είναι αυτά που λέτε και διαβάζοντας τα δημοσιεύματα στον τύπο, κάποιοι στη δική μου εκλογική περιφέρεια σκέφτονται ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέτε. Ε, ε επικοινωνιακό πρόβλημα έχετε μάλλον ε, μήπως πρέπει να καταργήσουμε κάποια προϊόντα. Λένε διάφοροι ότι πρέπει να καταργήσουμε κάποια είδη προϊόντων, παραγόγων. Ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν ναι, ακολουθήσει σχετική παγκόσμια νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή να καταργηθούν προϊόντα μεταξύ ε, ε, κάποια από τα οποία χρησιμοποιείτε κι εσείς. Τώρα, σε σχέση με αυτά που μας είπατε για την ε, κερδοσκοπία, μπορείτε να είστε λίγο ακριβέστερος. Ωραία, τι εστί η κερδοσκοπία. Μπορείτε εσείς να μας ορίσετε την κερδοσκοπία. Είναι απαραίτητα κακή η κερδοσκοπία. Λάγκεν Εγώ δεν έχω πρόβλημα να θέσει και άλλα ερωτήματα ο κύριο Ράτε Μάχερ αν το θέλει. Αλλά θα ήθελα από τη δική μου μεριά να πω και εγώ κάτι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε παρόν και έχετε εκφράσει τη θέση τη Goldman Sachs. Εγώ θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την ε, μορφή που θα πάρει το μέλλον. Ελέγχθη καταρχήν ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων τα οποία θα διαβιβαστούν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της ε, διαφάνειας. Αυτό είναι δύσκολο να το εξασφαλίσει κανείς. Εμείς λέμε ότι είναι ίσως υπερβολικό να έχουμε διαφάνεια σε όλα, αλλά αν δεν έχουμε αρκετή διαφάνεια δεν επιτυγχάνουμε το, το στόχο μας. Εδώ έχουμε από τη μία πλευρά τους Αμερικανούς οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο χώρο των ε, συναλλαγών εκεί. Η ευρωπαϊκή πλευρά θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να έχει και κάποια εποπτεία για αυτά τα οποία γίνονται στις αμερικανικές αγορές. Είναι γεγονό, είπατε ότι πράγματι είναι επικίνδυνο να συγκεντρώνονται όλα σε ένα φορέα. Για μένα θα ήταν μια πραγματική δοκιμασία αυτό το οποίο έγινε με την ε, Lehman Brothers. Αυτό κλειδώνησε το σύστημα και κινδύνευσε να υπάρξει μια κατάρρευση του συστήματος. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από τη δική σας πλευρά πώς το κρίνετε αυτό, πώς το σχολιάσετε. Το τρίτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε την ανάγκη να υπάρξει μια διαφορά σε κανονισμούς διαφάνειας μεταξύ της ε, συναλλαγών που αφορούν με επιχειρήσεις αφενός και συναλλαγών που αφορούν καθαρά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Όλη Σμιθ. Μήπως θεωρείτε ότι το σύστημα αμοιβών των στελεχών, το σύστημα των πριμ και των πόνους οδηγεί σε μια τάση να υποτιμούν ριζικά τους κινδύνους. Έχουμε δει τα τελευταία δέκα χρόνια ότι το τμήμα των χρηματοοικονομικών ε, ε, ε, υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μεταξύ 5 και 7% αλλά πήρε τα 40% περίπου των κερδών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως και το, το σύστημα αμοιβών παίζει κάποιο ρόλο. Η Goldman Sachs είναι μια επιτυχημένη εταιρεία η οποία έχει λειτουργήσει έτσι την αγορά παραγόγων ώστε να μην έχει καμία ευθύνη για τους κινδύνους στην αγορά αυτή. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε όλοι. Ότι η ελληνική κρίση δεν είναι απόλυτα απομονωμένη από την γενική κατάσταση της αγοράς. Και βλέπουμε και στην γερμανική ε, κοινή γνώμη να υπάρχει υπερβολική εστίαση στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος ακόμα και αν στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία προέρχονται από την ίδια την Ελλάδα, δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό καθαρά απομονωμένα, σαν να μην έχει σχέση με τίποτα άλλο. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε περισσότερο για την εποπτεία, για τι στατιστικέ, για τη διαφάνεια. Αλλά τι θα επιτύχουμε με όλα αυτά. Μπορούμε να περιγράψουμε τις διαδικασίες της αγοράς, αλλά δεν έχουμε βρει πραγματικά τι αιτίε όλων αυτών των φαινομένων. Μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα τι έχει γίνει, να έχουμε καλύτερη διάγνωση και ανάλυση. Αλλά αυτό δεν μα δείχνει ποιε είναι οι αιτίε των φαινομένων, ακόμα και ξέρουμε πώ λειτουργούν οι αγορέ. Επομένω, παραμένουμε σε ένα επίπεδο συμπτωματολογία. Εγώ νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και υπενθυμίσω αυτό που λέει η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ και υποδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αιτίες στην χρηματοοικονομική κρίση για το γεγονός ότι οι τράπεζες, οι κανονικές τράπεζες και οι τράπεζες επενδύσεων έχουν υπερβολική διασύνδεση μεταξύ τους και ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερος διαχωρισμός επενδυτικών τραπεζών και εμπορικών τραπεζών και βλέπουμε ότι στη Γερμανία οι τράπεζες ταμιευτηρίου και άλλες τράπεζες επλήγησαν από την κρίση παρά το γεγονός ότι δεν διαχειριζόντουσαν και δεν εμπορευόντουσαν επενδυτικά προϊόντα. Επίσης αναφέρθηκε τι τελευταίες, εβδομάδε ότι υπάρχει και μία ε, μεγάλη ανισότητα σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πλεόνασμα στο εμπορικό της ισογυζύγιο και αυτό μπορεί να έχει κάποιες ε, επιπτώσεις στην περίπτωση της ε, κρίσης στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω από εσά κάτι για αυτό το σημείο και αν αυτό είναι κάτι περαιτέρω πρέπει να εξετάσουμε. Νομίζω ότι προσπαθούμε τώρα να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Κύριε Κόργαν, αν θέλετε να πείτε κάτι για τα θέματα αυτά, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα προσπαθήσω να σταθώ σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα και θα τα παραπέμψω άλλα στον κύριο Μέτκαλφ. Είναι, λέτε ότι αυτά τα οποία λέω έχουν νόημα, αλλά κανείς δεν, δεν τα χάβει. Η κοινή γνώμη, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρώπη, εδώ στις Βρυξέλλες, οπουδήποτε. Είναι εξοργισμένη κοινή γνώμη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και έχουν το δικαίωμα να είναι εξοργισμένοι για αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους. Αλλά όλοι μας, ιδίως αυτοί που βρισκόμαστε στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχουμε μια πολύ βαριά ευθύνη για να προσπαθήσουμε να συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο που θα, είναι, θα βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει λίγο καλύτερα τι συμβαίνει και τι συνέβη. Πολλά πράγματα έγιναν στι ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν έρχονται από τι ΗΠΑ, οι οποίοι εμπλέκονται σε όλα αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εν μέρη απεδέχθη την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ με την ελπίδα ότι ίσως μπορώ να σας βοηθήσω λιγάκι στο να υπάρξει καλύτερη κατανόηση ορισμένων από αυτά τα θέματα και το τι πρέπει να κάνουμε για να μεταπίσουμε την κοινή γνώμη και να καταλάβει τι γίνεται. Επομένως κατανοώ απόλυτα αυτό το οποίο είπατε. Τώρα τι είναι προϊόντα χρηματοοικονομικά και πότε είναι προϊόντα απλώς και πότε φτάνουμε στην κερδοσκοπία. οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και εδώ ίσως, θα δεχόταν ίσως αυτό το οποίο είπα, ότι η κερδοσκοπία η οποία βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των ρυθμιστικών κανόνων είναι θετική. Γιατί χωρίς την κερδοσκοπία με την καλή έννοια της λέξης κερδοσκοπία είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά συστήματα. Κάποιος πρέπει να παίρνει κινδύνους. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικροί τραπεζίτες, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλες τράπεζες. Δεν θέλουμε να έχουμε μια κουλτούρα που λέμε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα με το, του κόσμου με το να απαγορεύουμε στον κόσμο να ρισκάρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει αρνητική βέβαια κερδοσκοπία. Είναι σαφές αυτό. Και το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αναφερόμενο στην πορνογραφία είπε ότι σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που ε, είναι πραγματικά αρνητική για όλο τον κόσμο και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την κερδοσκοπία, για την απαγόρευση των ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Νομίζω ότι η ίδια η αγορά τα καταφέρνει πολύ καλά. Όχι το, στο να απαγορεύει ορισμένα προϊόντα, αλλά να ξεφορτώνεται προϊόντα τα οποία είτε δεν λειτουργούν όπως προβλεπόταν να λειτουργήσουν ή έχουν στροβλε, στρεβλωτικά αποτελέσματα. Είναι σαν, σαν τα φάρμακα κατά κάποιο τρόπο, τη συνταγογράφηση φαρμάκων από τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα εξαφανίζονται. Στις πιο δύσκολες μέρες της κρίσης υπήρχαν ορισμένα υπερβολη... εξαιρετικά ε, δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα με πολλά ε, επίπεδα και ενσωματωμένη μόχλευση. Όλα αυτά όμως σε μεγάλο βαθμό εξαφανίστηκαν. Αυτό μπορεί να λυπεί ορισμένους αλλά αυτό σημαίνει ότι και αυτοί οι οποίοι πουλούσαν αυτά τα εργαλεία και αυτοί που τα αγοράζανε στο μέλλον θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί για να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα προϊόντα δεν θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα το αρνητικό που είχαν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ βρίσκω ότι είναι επικοδομητικό. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό δίνω κάποια απάντηση στο ερώτημά σας. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τον κίνδυνο σε σχέση με τις ίδιες τις ε, υποδομές του χρηματοοικονομικού συστήματος. Και επίσης αναφέρθηκε το θέμα της αμοιβή των στελέχων και των κινήτρων. Αυτό είναι ένα γενικό θέμα. Το Ένα σημαντικό λοιπόν θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπήρξανε κάποιες αστοχίες, κάποιες ε, ελλείψεις ισορροπίας μεταξύ, μέσα στην ισορροπία μεταξύ αμοιβών και ανάληψης κινδύνου. Υπήρξαν κάποιες επιχειρήσεις που δεν τα κατάφεραν πολύ καλά, αλλά μια εταιρεία όπως εμείς, η Goldman Sachs, καταφέραμε πολύ καλά να μην πέσουμε στη Λούμπα. Καταφέραμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά στα θέματα αυτά. Εξακολουθούμε να είμαστε μια, ε, μια ομόρφη εταιρεία ουσιαστικά. Και υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο αμοιβών των ανώτερων στελεχών που αποφασίζεται από τους εταίρους σε αυτή την ομόρφημη εταιρεία. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση που λαμβάνεται για την αμοιβή αυτών των στελεχών. Πληρώνονται καλά τα στελέχη της Goldman Sachs, αλλά έχουν μια δουλειά η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχουν οι περισσότεροι. Και το θέμα τώρα της ευθύνης των πολιτών, της διαχείρισης του κινδύνου, της αμοιβή και τον ΠΡΙΜ, αυτό είναι ένα θέμα δύσκολη ισορροπία. Το έχουμε το Χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουν πολύ. Και ένα τελευταίο θέμα και μετά θα κλείσω. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν μια σύγκριση ή μια καταναλογία αντιμετώπιση τραπεζών και επενδυτικών τραπεζών. Αν δείτε, άμα δείτε το παραδοσιακό γενικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας όπως λειτουργεί στην αγορά και της ε, εταιρείας holding στις Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν πάρα πολύ τελικά σε σχέση αυτές οι δομές σε σχέση με το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τις δυνατότητες που μπορούν να κάνουν. Η μόνη μεγάλη διαφορά είναι το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τράπεζες είναι κάπως απομονωμένες και δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αλλά αν δείτε μεγάλες τράπεζες και εταιρείε holding στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι αυτοί οι φορείς εμπλέκονται ιδιαίτερα και σε δραστηριότητες επενδυτικών τραπεζών, ώστε η ταμπέλα τράπεζα αφενός, επενδυτική τράπεζα αφετέρου, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα στην πράξη. Κύριος Μέρκαλ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λάγκεν, νομίζω πως ε, αναφέρατε κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται με υποδομή, με την υποδομή. Λυπούμε λοιπόν, αν δεν ήμουν ε, σαφής όσον αφορά το θέμα της εμπιστευτικότητας. Εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο είναι σημαντικό, αλλά είναι και επίγον να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σε όλες τις δικαιοδοσίες. Όμως, επειδή η βασική πρόκληση με το εμπορικό αρχείο είναι να είναι παγκόσμιο, Πολύ γρήγορα προσκρούμε σε προβλήματα όπως πάμε σε μια δικαιοδοσία, πάμε σε μια άλλη ε, δικαιοδοσία όπου οι επόπτες μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν είναι τώρα ίσως σωστό να μπούμε σε λεπτομέρειες για τη δουλειά που κάνουμε, αλλά ευχαριστώ θα μπορούσα διμερώς ή με οποιαδήποτε ομάδα βουλευτών να έρθω και να σας πω λεπτομερώς τι ακριβώς κάνουμε, με ποιους συνεργαζόμαστε στο μέτωπο τη εποπτείας. Ευχαριστώ μπορούμε να σα δώσουμε τα στοιχεία γιατί είναι προ το δικό μα συμφέρον ώστε οι επόπτες να μπορέσουν ακριβώς να φτιάξουν αυτή την ακριβή και κέρια εικόνα για την ανακατανομή του κινδύνου εντός της αγοράς. Αυτό μας οδηγεί στο άλλο ερώτημα της πρόσβασης που δεν είναι διόλου ε, μικρότερη σημασίας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή τη βασική αρχή της πρόσβασης ώστε να το ενθαρρύνουμε. Αλλά δεν είναι απόλυτα στο δικό μας έλεγχο. Είναι ωστόσο ενθαρρυντικό ότι τα υπάρχοντα μητρώα συναλλαγών συνεργάζονται όχι μόνο με τους υπόπτους αλλά και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς από όσο γνωρίζω. Και η ομάδα διεθνών αριθμιστών εργάζεται για, μια ολόκληρη σειρά, για ένα πρωτόκολλο ώστε να διασφαλίσει πως ε, ο χειρισμός της πρόσβαση θα γίνει με ταχύ και καλά οργανωμένο τρόπο στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει εδώ βάση, υπάρχει, ε, βάση για αισιοδοξία σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και όσους έμειναν θέλει ποιος να κάνει κάποια τελική παρέμβαση. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν πιστεύετε πως έχετε κάτι να πείτε που δεν το είπατε ακόμα, ευχαρίστω. Θέλετε κύριε Μέρκαλφ να πείτε κάτι τελευταίο. Τέλος, ναι, ένα σύντομο σχόλιο που σχετίζεται με την απαγόρευση προϊόντων. Νομίζω πως είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και να θυμόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκαν οι αγορές παραγόγων ήταν ως απάντηση στον αυξημένο κίνδυνο αυτή ήταν η βασική όθηση και αυτό δείχνει ο χρόνος κατά τον οποίο αυτά όλα έχουν αναπτυχθεί. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, το να απαγορεύσουμε τα παράγωγα δεν θα έλυνε το υποσκάπτον πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε κύριε Κόργαν και κύριε Μέτ Metcalf για τις, την απόπειρά σας να απαντήσετε σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα ερωτήματα. Το ξέρω ήταν δύσκολο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σε αυτήν την ακρόαση. Ε, Συμβάλλατε όχι μόνο για την εξέταση του θέματος που είχαμε επιτάπητος, αλλά και για τα μελλοντικά και όσοι έμειναν σίγουρα θα σας εκτίμησαν την παρέα της παρεμβάσης σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, and, and Επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται για τις 19 Απριλίου στο Στρασβούργο στις 7 με 8.30 το βράδυ. Σας ευχαριστώ. Πέρα συνεδρίασης.